Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you at this important meeting of the COCOBU. I have to apologize that uh, we started a bit too late. In my agenda, another room was indicated. And... Έγινε μικρό μπέρδα με την αίθουσα που θα κάναμε την ε, συνεδρίαση. Τέλος πάντων, λυπάμαι για τον μπλέξιμο που έγινε όσον αφορά αυτή την τη συνεδρίαση και τέλο πάντων είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή συνάντηση, διότι πρόκειται να έρθει εδώ ο πρόεδρο του Ελληνικού Συνεδρίου για να μα παρουσιάσει ε, την εισήγησή του και έχουμε επίση και άλλα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου που παρίστανται εδώ και φαντάζομαι ότι όλοι έχετε λάβει την ε, ημερησία διάταξη και θέλω να μου πείτε αν έχετε τίποτε παρατηρήσει επί τη ημερησία διατάξεω. Εάν όχι, τότε θεωρώ ότι εγκρίνεται την ημερησία διάταξη και θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη σας ότι μεταδίδεται μέσω ίντερνετ αυτή η συνεδρίαση. Οπότε ό,τι λέτε, ό,τι λέτε είναι κοινό κτήμα. Άρα θα πρέπει να έχετε μέσα στις κάρτες ψηφοφορίας μια που θα ψηφίσουμε. Όποιος δεν τις έχει ας πάει τις βρει. για να εγκρίνουμε τώρα ε, τα πρακτικά των προηγουμένων μας συνεδριάσεων. Όχι από ό,τι βλέπω, επομένως ε, δεν υπάρχει καμία ένσταση. Θεωρώ εγκεκριμένα τα πρακτικά. Πάμε στο σημείο 4 της μερικής διατάξεως. Είναι το πιο βασικό θέμα της σημερινής διατάξεως και είναι η σύγκριση και παρουσίαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Νεκτικού Συνεδρίου της ετησίας εκθέσεως για τη χρήση του 2010. Κύριε Καλτέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή για μένα σήμερα να σας παρουσιάσω για άλλη μια φορά την ετησία μας έκθεση όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού για τη χρήση 2010. Καθώς και την έκθεση για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης για το ίδιο οικονομικό έτος όπως και στο παρελθόν η τύση έκθεση για την εκτέλεση του προβλημού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως καλύπτει την αξιοπιστία των λογαριασμών και την κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων. Φέτος, η έκθεση επίσης περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο σχετικό με τα αποτελέσματα των δαπανών της ΕΕ. Η ποιότητα της έκθεσης είναι θέμα που επίσης το εξετάζουμε. Αφού σα παρουσιάσω τα βασικότερα μηνύματα, θα σα επισημάνω και κάποια άλλα συναφή ζητήματα. Αυτά προέκυψαν από τη μεταρρύθμιση του προπολογισμού και από τι εξελίξει στον τομέα τη οικονομική διακυβέρνηση. Όσον αφορά την αξιοπιστία των οργανισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το συνέδριο καταλήγει στο τηλεογραφισμό του 2010. Ακριβωδίκη εικόνα παρουσιάζουν για την οικονομική κατάσταση. Για πράξει, ταμιακέ ζωέ για αυτή την χρονιά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει περιθώριο βελτίωση για τα στήματα πληροφόρηση και την πληροφόρηση, κυρίω για να έχουμε καλύτερα στοιχεία για τους κινδύνου ει βάρο τη διαχείρισης. Φέρει πριν Το συνέδριο επισημαίνει ότι οι λογιστικοί κανόνες και η υποπτία δεν προσαρμόστηκαν όπω πρέπει για να επιχούν τη σημαντική αύξηση των προπληρωμών. Προχρηματοδότηση στον προπολογισμό Από το 2009 και μετά έχουμε σημαντική αύξηση πληρωμών. Συνεισφέρουν σε ταμεία με τα οποία εφαρμόζονται τα μέτρα χρηματοοικονομικής τεχνική στον τομέα τη συνοχή. Σύμφωνα με τα μέσα αυτά, ο προπολογισμό καλύπτει τι προπληρωμέ. Μόλι υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Τα κράτη-μέλη παραπέρα χρησιμοποιούν αυτά τα ταμεία και του πόρου για να παράσχουν ενισχύσεις, δάνεια, εγγύσεις, επενδύσεις για αυτόν τον προγραμματισμό. Και βρήκαμε ένα σωρό περιπτώσεις. Οπότε η Επιτροπή καταρχήν είχε καταχωρήσει τις πληρωμές αυτές στον προπολογισμό σαν δαπάνες και όχι ως ενεργητικό. Και γι' αυτό και οι προσωρινοί λογαριασμοί δίνανε την εντύπωση την εξή, ότι οι αποδείκτες των ενισχύσεων είχαν αιτιολογήσει την χρηματοδότηση. Όμως, στην πραγματικότητα, δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Οπότε και σε να έχουμε κινδύνους. Η Επιτροπή διόρθωσε τις ανακρίβειες. Προσαρμόσε τους λογαριασμούς. Και αναθεώρησε αυτά τα αντίστοιχα στοιχεία του λογαριασμού του 2009. Οπότε και επισύρουμε την προσοχή σας ή στο θέμα αυτό, στα πλαίσια της δήλωσης αξιοπιστίας στην αρχή τη έκθεση. Όμως, αυτό το ζήτημα δεν είναι θέμα μόνο λογιστικής. Διότι, βασικά, το θέμα είναι να δούμε πώ θα υπάρχουν αρκετέ πληροφορίε για διαχείριση, εποπτείας και διαχείρισης. Και γι' αυτό το συνέδριο πιστεύει ότι Επιγόντω θα πρέπει η Επιτροπή να, να θεωρήσει αυτόν τον κανόνα και θα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρο τόσο ώστε να εξασφαλίσει ότι οι απαραίτητε πληροφορίε είναι διαθέσιμε για τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να βελτιωθεί η υποπτία αυτών των μέσων ε, χρηματοοικονομική τεχνική. Και ε, από ό,τι γνωρίζω, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει μια πρόταση για τροποποίηση αυτών των σχετικών κανόνων. Και από ό,τι γνωρίζω, αυτά θα τα συζητήσετε εσεί σήμερα. Το βασικό μέρος τώρα των θεμάτων της ετήσιας έκθεσης και δύο εξοπιστίας αφορά την κανονικότητα για έσοδα και δαπάνες. Η ιδίωση εξοπιστίας το οικονομικό του 2010 έχει αναθεωρηθεί. Έτσι θα λάβουμε υπόψη τις ε, τροποποίησεις όσον αφορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα οποία τέθηκαν σε σχέση το 2011. Έχουμε επομένω πλέον διάκριση μεταξύ εσόδων, αναλήψεων, πληρωμών και υποχρεώσεων. Κατηνών του συνεδρίου. Τα υποκείμενα λογαριασμού έσοδα είναι νόμιμα και κανονικά. Το ίδιο και οι υποχρεώσει επίσης είναι νόμιμες και κανονικές. Όμως, όμως αντίθετα, οι πληρωμές έχουν σημαντικά σφάλματα. Και το σφάλμα πάει στο 3,7%. Σημειωτών, αυτό δεν αποτελεί θέμα περιπτώσεων απάντηση. Γιατί έχουμε πολλούς λόγους για τα σφάλματα και γενικά είδαμε ότι τα συστήματα ελέγχου ήταν εν μέρει αποτελεσματικά όσον αφορά την κανονικότητα. Για τις πληρωμές έχουμε ειδικέ εκτιμήσεις πέντε ομάδων τομέων πολιτικής. Αυτά τα αναφέρουμε στα κεφάλαια 3 έως 7 της έκθεσης. Αυτά αντιστοιχούν γενικά στην περίοδο 2007-2013. Και έχουμε περάσει κάποιες μεταβολές σε σχέση με προηγούμενες αιτήσεις εκθέσεις. Και έτσι θα έχουμε χρησιμότερη ανάλυση για τις δαπάνες. Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται στα αποτελέσματα δοκιμαστικών ελέγχων, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και εξέταση της αξιοπιστίας. Όπως παρουσιάζονται αυτά στην ετήσια έκθεση. Και τις εκθέσεις συγκεκριμένα των γενικών διευθύνσεων. Οπότε λέμε ότι δύο, μεγάλες, ε, δύο μεγάλοι τομείς πολιτικής, γεωργία δηλαδή και συνοχή, έχουν σημαντικά σφάλματα. Επομένω, τα συστήματα ελέγχου είναι εν μέρει αποτελεσματικά και γι' αυτό και η πολιτική συνοχή ε, ήταν τελικά ο τομέας των μεγαλύτερα λάθη. Πάμε στο 7,7% του 2010. Το ποσοστό αυτό είναι ψηλότερο από αυτά που είχαμε εκτιμήσει για τι δαπάνε του 2009 και αυτό εξηγεί την αύξηση στο σφάλμα σε σύγκριση με το παρελθόν για το σύνολο του προπολογισμού. Πάντως όπως και πέρυσι σας είπα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πριν εξαγάγουμε πια από τα συμπεράσματα. Γι' αυτό οφείλεται στο ότι είναι πολιετής αυτές οι δαπάνε και τα μέτρα. Και από χρονιά σε χρονιά αλλάζουν πληρωμές. Παρ' όλα αυτά, σχεδόν μισές του πληρωμές που πέρασαν από τον έλεγχο είχε σφάλματα. Τα σφάλματα κυρίως προέρχονται από σχετικά λίγα έργα μη επιλέξιμα και παραβιάσεις νομοθεσίας για τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του δημοσίου. Οπότε γι' αυτό και θεωρεί το συνέδριο ότι οι αρχές των κρατών μελών είχαν αρκετά στοιχεία και μπορούσαν να βρουν και να διορθώσουν τουλάχιστον κάποια από τα σφάλματα πριν τις πληρωμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαίνει πρόοδο σε σχέση με τις προηγούμενες μας συστάσεις. Όμω θεωρούμε ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο βελτίωση από των κρατών μελών για του μηχανισμού βελτίωση για τι δραστηριότητε. Και για αυτό υποβάλλουμε και περαιτέρω συστάσει. Όσον αφορά τη γεωργία και φυσικού πόρου, το σφάλμα πήγε στο 2,3%. Εν μέρει αποτελεσματικά τα συγκεκριτικά συστήματα. Οι άμεσες πληρωμές από το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης είναι αντίστοιχο 40 δισεκατομμυρίων από τα 57. Εκεί δεν είχαμε ουσιώδη σφάλματα. Όμως, η ορδική ανάπτυξη είχε σφάλματα. Διαπιστώσαμε ψηλή συχνότητα εμφάνιση φαλμάτων Λόγω του ότι ήταν απαρχαιωμένες οι βάσεις δεδομένων για τα χωράφια, για τις γεωργικές εκτάσεις, αυτά τα οποία ήλεγχαν εθνικοί επιθεωρητές, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία και κάτω χώρες. Έχουμε επίσης και κάποιες συστάσεις που τις ε, περιέχει η έκθεσή μας. Όσον αφορά τι δύο ομάδε του τομέα πολιτική έρευνα και τι λοιπέ εσωτερικέ πολιτικέ και εξωτερική βοήθεια και ανάπτυξη και διεύρυνση, το συνέδριο συνεπέρανε ότι συνολικά οι πράξει αυτέ δεν περιέχουν σιώδη σφάλματα. Όμω, τα συστήματα είναι μερίμοτα αποτελεσματικά και επίση έχουμε ακόμα κίνδυνο σφάλματο για τι ενδιάμεσε και τελικέ πληρωμέ. Εκεί είχαμε σφάλματα σημαντικά. εξωτερική βοήθεια επίση μέσω Ταμείου Ανάπτυξη. Έχουμε για, για αυτά σχετική χωριστή έκθεση και για το 2010 διαπιστώσαμε ότι οι πληρωμέ είχαν σφάλμα 3,4% και τα συστήματα ήταν μέρα αποτελεσματικά και για την τελική, τελευταία ομάδα πολιτικής, διοικητικέ και λοιπέ δαπάνε, καταλήξαμε ότι δεν είχαμε σφάλματα. Εδώ τα συστήματα είναι αποτελεσματικά όπως και στο παρελθόν. Συνολικά, ο έλεγχος για το 2010 μας ε, δικαίωσε όσον αφορά αυτά που είχαμε πει τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζουμε να έχουμε κάποιους κινδύνους για την κανονικότητα, για τους δικαιούχους, για διαρθρωτικές πολιτικές και για ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές. Όμω έχουμε βελτιώσει για αποτελεσματικότητα των συστημάτων. Σε επιτροπής και στη Γεωργία. Είχαμε ταυτόχρονα πρωτοτική τάση όσον αφορά το σφάλμα για τον προπολογισμό. Από το 7% συν του 2006 πήγαμε σε λιγότερο από 4% για το 10%. Επομένως, πώς συγκρίνονται η έλεγχη του συνεδρίου με τις επιτροπές, οι αιτήσει εκθέσεις γενικών διευθύνσεων και η συνθετική έκθεση της Κομισιόν περιέχουν πολλές επιφυλάξεις για τον εσωτερικό έλεγχο ο, για την κανονικότητα δαπανών στις διαφορετικές πολιτικές. Γενικά αυτές οι επιφυλάξεις πηγάζουν από τον υπολογισμό κινδύνου εισφάλματος. Μια που έλεγχος πάει για το όριο του 2% σε πολιτική βάση. Αυτό είναι στοιχείο για την αξιολόγηση. Όλο ένα και πιο σημαντικό για το 2010. Θα μπορούσε η Επιτροπή να ωφεληθεί αν αυτό το έκαναν με μεγαλύτερη συνέπεια όλες οι γενικές διευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, το συνέδριο βλέπει ότι όλες αυτές οι επιφυλάξεις θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες και για τη συνοχή. Επ' αυτού, το συνέδριο θεωρεί ότι η προσέγγιση της Επιτροπής μπορεί να οδηγήσει σε υποτίμηση του κινδύνου. Γι' αυτό και εμείς εμένουμε στις προηγούμενες παρατηρήσεις ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ποιότητα πληροφοριών για διορθώσεις και ανακτήσεις. και οι αιτήσει εκθέσει των διευθύνσεων επίσης αξιολογούν επιδόσει και φέτο για πρώτη φορά στο κεφάλαιο 8 της έκθεση, το συνέδριο παρουσιάζει εξετάσεις, συγκρισιμότητα και αξιοπιστία όλων αυτών των ε, πληροφοριών από Γενικές Διευθύνσεις, Γεωργίας, Γεωργικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Πολιτικής, Έρευνας και Καινοτομίας. Αυτά είναι η βάση για να συστήσουμε να επικεντρώνει την Επιτροπή περισσότερο στα, στις εκθέσεις δραστηριοτήτων. Οικονομία, αποδοτικότητα των χρηματοδοτήσεων. Να έχουμε στόχους ενδιάμεσους για τους πολιτείς στόχους και έτσι να βλέπουμε αν υπάρχει πρόοδος. Η καλή ποιότητα είναι το κλειδί για να έχουμε λογοδοσία των υπεύθυνων της διαχείρισης. Στο κεφάλαιο 8 επίσης έχουμε και άλλες συστάσεις για τον έλεγχο της επίδοσης για, το, για την προηγούμενη χρήση όπως τα είπαμε στις εκθέσεις του συνεδρίου και συγκεκριμένα στην συνδιαχείριση συστήνουμε τρία τεινά προς την Επιτροπή για να έχουμε καλύτερη ποιότητα των στοιχείων. Πρώτον, περισσότερη προσοχή στο σχεδιασμό για τις δαπάνες και να καθοριστούν οι κίνδυνοι κατά την υλοποίηση. Δεύτερον, δεύτερον συνεπείς δείκτες επιδόσεων, αξιοπιστία πληροφοριών για στόχους και αποτελέσματα και τρίτον, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν συστήματα παρακολούθηση και έτσι να ξέρουν τι γίνεται με τα στοιχεία και τα αποτελέσματα. Αυτέ οι συστάσει, Πρόεδρε, Επίση μπορεί να είναι εσεί στην Επιτροπή. Για ανάπτυξη έκθεση αξιολόγηση στο πλαίσιο δικασία απαλλαγή, όπω τα αναφέρει το άρθρο 319 τη νίκη τη Λισαβόνα. Όντω, Πρόεδρε, αυτά έχουμε να πούμε. Όσον αφορά τη σύνοψη των όσων αναφέρει η έκθεση για τη χρήση 2010 και πιστεύω ότι έτσι επιβεβαιώνεται το βασικό μήνυμα των προηγουμένων χρήσεων παρά τις ε, βελτιώσεις των συστημάτων έχουμε ακόμα κινδύνους για την κανονικότητα. Αντιμετωπίζονται μόνο με μεταρρύθμιση νομοθετικού πλαισίου και επανασχεδιασμό συστημάτων ελέγχου. Και οι προτάσεις για δαπάνη το 2004 θα είναι η ευκαιρία. Όμως όπως τόνισα και πέρσι, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αφορούν τη βελτίωση γενικώ των δαπανών για τη διαχείριση, περιορισμό κινδύνων, για κανονικότητα και επιδόσεις και μείωση του κόστους των ελέγχων επίσης. Χρειάζονται κατάλληλες ρυθμίσεις για να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και λογοδοσία. Και αυτό είναι η πρόκληση μεγάλη. Όπως λέει η έκθεση, χρειάζεται να καθοριστούν σαφείς στόχοι. Να βελτιωθούν τα συστήματα για να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία για πρόοδο και κινδύνους και πέρα από αυτές τις νέες προτάσεις που αφορούν τον προπολογισμό έχουμε σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Εδώ έχουμε σημαντικά ζητήματα διαφάνειας και αυξάνουμε τα κενά στη λογοδοσία και δημοσιονομικό έλεγχο. Αυτά τα τόνισε η Επιτροπή Επαφής. των οργάνων ελέγχου. Είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, λογοδοσία και έλεγχος όποτε έχουμε να κάνουμε με δημόσιες δαπάνες. Και γι' αυτό και θεωρείται αυτό μια ευκαιρία, ούτως ώστε αυτέ οι αρχέ να υλοποιηθούν κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι βουλευτές. Όταν διακυβεύονται δημόσια κονδύλια, οι πολίτες έχουν θεμητή προσδοκία. Οι ελεγκτές έχουν αποτελεσματικό έλεγχο και λογοδεσία. Και είμαι βέβαιος ότι η ετησία έκθεση που είχα την τιμή να σα παρουσιάσω σήμερα θα σας δώσει μία στέρεα βάση ούτως ώστε όλα όσα επιθυμούν για τα κονδύλια της Ένωσης για τη Χρήση του 2010 να ευοδοθούν. Διαφάνεια και λογοδοσία. Είναι ευθύνη όλων μας στη μια δημοκρατική κοινωνία και κυρίως υπό την σημερινή συγκυρία που η πίεση είναι σημαντική. Η σημασία επομένω να πετύχει έψον του στόχου τη είναι πάρα πολύ μεγάλη και έτσι θα πρέπει επομένω να αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Και σα ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Καλδέιρα, η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου παρακολουθείτε από τα μέλη της ε, Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου μεγάλη προσοχή. Και σίγουρα και σε αυτή την περίπτωση θα ελέγξουμε την εκθεσή σας με μεγάλη προσοχή. Ο τελικός αποδέκτης της ε, έκθεσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την καλωσορίζω και θέλω να της δώσω το λόγο για να ακούσουμε τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα όσα είπε ο κ. Σκαλδέιρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγητά, αγαπητοί βουλευτές της ε, Επιτροπής αυτής και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2010 μαζί με τις απαντήσεις της Κομισιόν είναι το αποτέλεσμα μιας εντατικής και επικοδομητικής συζήτησης μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας η διαδικασία κινείται πιο ομαλά. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τον πρόεδρο Καλνταΐρα, τα, μέλη, του ελεγκτικού συνεδρίου και τις υπηρεσίες για τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε. Η έκθεση δημοσιεύεται σε μια χρονική στιγμή όπου συμβαίνουν κρίσιμες αλλαγές και στην οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη μελλοντική διαχείριση του προϋπολογισμού της. Οι συζητήσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο οι κανονισμοί και ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός είναι πολύ σημαντικοί για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Είναι ακόμα πιο σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο να έχουμε ε, κριτήρια σταθερά, σαφή, όπου οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη μπορούν να βασίζονται σε αυτά. Και με βάση αυτά να προσμετρούμε τα λάθη. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν σταθερή και αξιόπιστη πληροφορία για τα λάθη, τις δαπάνες, τα διορθωτικά μέτρα, ούτω ώστε να μετρήσουμε την πρόοδο που σημειώνεται συν το χρόνο. Η σωστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών απαιτεί σοβαρή διαχείριση και σοβαρό σύστημα ελέγχου. Η Κομισιόν ακριβώς έκανε προτάσεις στον αθωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό προς αυτή την κατεύθυνση, ούτω ώστε να έχουμε έναν έλεγχο αποτελεσματικό ε, και μια διαχείριση αποτελεσματική, ειδικά στους τομείς που υπάρχει μεικτή ευθύνη για τη διαχείριση. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα βασικά μηνύματα της ετήσιας έκθεσης ε, του κ. Καλντέιρα. Σε ό,τι αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς, το συνέδριο για τέταρτη συνεχή χρονιά έχει εκδώσει μια θετική γνωμοδότηση. Χαίρομαι που οι προσπάθειές μας ε, οδήγησαν σε αυτή την θετική αξιολόγηση από το ελεκτικό συνέδριο. Παρ' όλα αυτά, το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι δεν υπάρχει συστηματικός συμψηφισμός της προχρηματοδότησης. Η Κομισιόν ε, πρότεινε να υπάρξει μια διάταξη στο δημοσιονομικό κανονισμό, ούτως ώστε να υπάρχει ε, υποχρεωτικός συμψηφισμός αυτών των πληρωμών. Ε, βασιζόμαστε στους συνομοθέτες για να μας υποστηρίξετε, στο Κοινοβούλιο δηλαδή. Το συνέδριο επίσης θεωρεί ότι κάποιες πληρωμές που γίνονται από τις εθνικές αρχές με βάση τα μέσα οικονομικής ε, τεχνικής πρέπει να θεωρηθούν ως μεταφορές ε, προσόδων και όχι ως δαπάνες. Για το 2010 αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε μετά από την επίκληση της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη να δώσουν τα απαραίτητα ε, στοιχεία ε, σε εθελοντική βάση. Η Κομισιόν επίσης ε, πρότεινε να βελτιωθεί η τρέχουσα νομική βάση, ούτω ώστε να έχουμε συστηματικά από τις εθνικές αρχές τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να κάνουμε σωστούς λογαριασμούς. Επίσης, αυτό θα βοηθήσει να υπάρχει σωστή παρακολούθηση από τις, από τις αρχές διαχείρισης στα κράτη-μέλη. Το 2010 το ποσά προχρηματοδότησης έφτασαν στα 54,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ συμπεριλαμβάνουμε και την, ε, την προσαρμογή των 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν τα μέσα ε, οικονομικής τεχνικής, χρηματοοικονομικής τεχνικής. Όπως είπα και νωρίτερα, η Κομισιόν θα το παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς αυτό το θέμα ε, από την πλευρά της διαχείρισης και της λογιστικής. Το 2010 το πλεόνασμα του προϋπολογισμού έφτασε τα 4,55 δις ευρώ και καλύπτει και τις δαπάνες αυτό το ποσό και τα έσοδα. Αυτή η αύξηση οφείλεται στο ότι η Δημοσιονομική Αρχή δεν ενέκρινε το συνήθι τροποποιητικό ε, προϋπολογισμό που η Κομισιόν προτείνει στο τέλος του χρόνου. Η αύξηση όμως στο πλεόνασμα πρέπει να συνδεθεί και με την υποεφαρμογή σε πολλούς τομείς που φτάνει τα 2,73 δισεκατομμύρια ευρώ υπό εφαρμογή των δαπανών. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως σε μια πιο ε, στεναρή προληπτική στάση που τηρεί η Κομισιόν. Τα πιο σημαντικά ποσά προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπου η Κομισιόν ακολουθεί μια αυστηρή πολιτική διακοπής και αναστολής των πληρωμών. Σε ό,τι αφορά την νομιμότητα και τακτικότητα των συναλλαγών, ε, έχουμε παραμείνει σχεδόν στο status quo. Θα ήθελα να αναγνωρίσω σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορους τομείς και τη συνέχιση της ε, θετικής αυτής τάσης της περασμένης χρονιάς εκτός από την πολιτική συνοχής. Καταρχάς, από πέρυσι ε, το πιθανό ποσοστό σφάλματος για όλες τις ε, ευρωπαϊκές δαπάνες βρίσκεται εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το 4%. Αυτό σημαίνει ότι η ευρεία πλειοψηφία πάνω από 96% των συνολικών πληρωμών που έγιναν το 2010 δεν είναι εντελώ αλάνθαστες. Επιπλέον, όλες οι δεσμεύσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής και τα έσοδα για τον συνολικό ενωσιακό προϋπολογισμό δεν είχαν λάθη. Δεύτερον, έχουμε θετικά αποτελέσματα για πολιτικές που διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τομείς όπως η έρευνα και άλλες εσωτερικές πολιτικές, η εξωτερική βοήθεια, η αναπτυξιακή βοήθεια, η διεύρυνση και οι διοικητικές δαπάνες όλο και βελτιώνονται. Το ποσοστό σφάλματος για τα σχετικά κεφάλαια στην έκθεση του συνεδρίου ε, είναι κάτω από το κατόφλι σημασίας. Τρίτον, η κατάσταση στη γεωργία παραμένει σταθερή με ένα επίπεδο λάθους κοντά στο κατόφλι του 2%. Επίσης, το 2010 το συνέδριο επιβεβαιώνει ότι οι πληρωμές για τις άμεσες ε, επιδοτήσεις σε εκατομμύρια αγρότες που είναι περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έφεραν, ήταν αλάνθαστες. Ε, σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχής, το, δυστυχώς το σφάλμα ε, αυξήθηκε ε, σε σχέση με το 2009, αλλά παρόλα αυτά βρίσκεται αρκετά κάτω από τα επίπεδα που είχαμε το 2006, το 2007 και το 2008. Αυτό, αυτή η αύξηση οφείλεται στον κύκλο ε, δαπανό ε, στην πολιτική συνοχή. Τα περισσότερα προγράμματα ξεκίνησαν πέρυσι, τα παρελθόντα χρόνια μάλλον, και πληρώνονται από το 2010 και μετά. Το ποσό των διάμεσων και τελικών πληρωμών ουσιαστικά διπλασιάστηκε. Όμως οι βασικές πηγές φάλματος οφείλονται κυρίως στα, στους πιο περίπλοκους κανόνες επιλεξιμότητας ε, που αφορούν τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές. Από την άλλη, οφείλεται σε αδυναμίες, σε ορισμένα συστήματα κρατών μελών, περιορισμένα όμως, ε, και που αφορούν όμως λίγα προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν εστιάζει την ενίσχυσή της ε, και ενισχύει την εποπτεία της σε αυτούς τους πιο ασθενείς κρίκους. Ο στόχος είναι διτός. Καταρχάς, να υποστηρίξουμε την προσπάθεια ε, όλων αυτών που πρέπει να βελτιώσουν τα συστήματά τους και δεύτερον, όπου δει, θα πρέπει να έχουμε προληπτικούς μηχανισμούς διακοπή και αναστολή των πληρωμών, δηλαδή αν χρειάζεται για να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το 2010 η Κομισιόν κατ' επανάληψη χρησιμοποίησε τα μέτρα, τα προληπτικά και τα διορθωτικά που έχει στη διάθεσή τη. Φερρυπίν, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Κομισιόν διέκοψε τις πληρωμές ε, ύψους 2,15 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη-μέλη και συγκεκριμένα στις διαχειριστικέ αρχές των κρατών μελών. Το σχετικό ποσό για το Κοινωνικό Ταμείο ήταν 255 ε, εκατομμύρια. Η, Αρχέ διαχείρισης στα κράτη-μέλη είναι υποχρεωτικές να λογοδοτούν και αυτό ξεκίνησε υποχρεωτικά να ισχύει από το τέλος του 2010. Η Κομισιόν εκτιμάει ότι αυτή η νέα υποχρέωση θα δώσει περισσότερες πληροφορίε και διασφάλιση σε ό,τι αφορά τον τρόπο που οι εθνικές αρχές εφαρμόζουν τα προγράμματα της πολιτική συνοχή στη σημερινή περίοδο προγραμματισμού. Η Κομισιόν θέλει να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσει τη διαχείριση των ε, ταμείων στην επόμενη γενιά προγραμμάτων. Ακριβώς γι' αυτό πρότεινε να βασίσει τη σχέση της με τα κράτη-μέλη σε, σε συμβόλαια εταιρική σχέση, Συμβάσει εταιρικέ σχέσει. Και η Κομισιόν θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ πώ ε, επιτυγχάνουν του στόχου τα κράτη-μέλη την αιρεσιμότητα, την επιλεξιμότητα που ε, υπάρχουν σε αυτές τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης. Η Κομισιόν προτείνει και ένα νέο πλαίσιο ελέγχου που θα βασίζεται σε ελεγχόμενους ετήσιους λογαριασμούς που θα λάβει διασφάλιση διασφάλιση από τις ε, εθνικές διαχειριστικές αρχές κάθε χρόνο. Τα κράτη-μέλη θα χάσουν ουσιαστικά τμήμα των ε, οριστικά τμήμα των κοινοτικών κονδυλίων, εάν τα συστήματά τους δεν ανοιχνεύουν τις παρατυπίες πριν υποβάλουν ε, τις αιτήσει για αποζημίωση ε, προς την Κομισιόν. Θέλω να υπενθυμίσω ότι λάθος δεν σημαίνει απάτη. Το ότι συμβαίνει δεν σημαίνει ότι τα κονδύλια έχουν εξαφανιστεί, έχουν σπαταληθεί. Σημαίνει ότι κάποια σχέδια, κάποια προγράμματα είχαν αδυναμίες στην εφαρμογή τους, όπως ε, σε ό,τι αφορά τη δήλωση των ε, μη επιλέξιμων δαπανών ή λάθη στον υπολογισμό των δαπανών. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ειδικοί και σε εκθέσεις του ελεκτικού συνοδρίου είναι μια πολύτιμη συνεισφορά. Γιατί ε, οθούν σε περισσότερε ε, βελτιώσει ε, με σε ό,τι αφορά τον τρόπο που οι υπηρεσίε τη Κομισιόν και άλλοι φορεί παρακολουθούν τα προγράμματα και αυτέ οι χρηματοδοτούμες δραστηριότητες έχουν προσθέμενη αξία. Ε, στην ανακοίνωση που υιοθέτησε τον Ιούνιο αυτή η Κομισιόν για το πολιτέ πρόγραμμα ε, τόνισε την προτεραιότητα που δίνει σε, στην επόμενη γενιά προγραμμάτων σε μια προσέγγιση που θα πετυχαίνει τους στόχους. Εντοπίζουμε στόχους, ε, ορόσημα, ε, επιδόσεις, δείκτες επιδόσεων ε, σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις. Μέχρι το τέλος του χρόνου η Κομισιόν επίσης θα εκδώσει την πρώτη έκθεση αξιολόγησης που θα βασίζεται στο άρθρο 318 της Συνθήκης. Αγαπητοί βουλευτές της Επιτροπής αυτής και του Ελεκτικού Συνεδρίου, Είμαι πολύ ικανοποιημένο που το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο επιβεβαιώνει ότι η Κομισιόν είναι στο σωστό δρόμο, σωστή πορεία. Η Κομισιόν γνωρίζει το, τα σημερινά προβλήματα και αναλαμβάνει πλήρω την ευθύνη για να αντιμετωπίσει του τομεί όπου χρειάζονται βελτιώσει. Ξέρουμε ότι χρειάζονται περισσότερε προσπάθειε και ότι αυτέ οι προσπάθειε θα πρέπει να γίνουν από όλου του οικονομικού φορεί και κυρίω από τι εθνικέ αρχέ διάφορα νέα μέτρα που περιλαμβάνουν τις προτάσεις μας για την επόμενη περίοδο δαπανών, ε, την επόμενη γενιά, ε, υπάρχουν ε, και προτείνονται, έχουμε πνευστεί από τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου και από την αρχή απαλλαγής οι προτάσεις μας δείχνουν ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη απλούστευση, διαφάνεια, μεγαλύτερη λογοδοσία από όλους τους οικονομικούς φορείς και μηχανισμοί ελέγχου αποτελεσματικοί σε σχέση με το κόστος τους. Τώρα, αν αυτά τα μέτρα θα γίνουν ε, ενωσιακό δίκαιο, αυτό εξαρτάται κυρίως από τους συνομοθέτες. Η θέση της Κομισιόν παρουσιάζεται πλήρως στις προτάσεις της και η δέσμευσή της να βελτιώσει περαιτέρω την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους επόμενους μήνες, διάφοροι συναδελφοί μου και εγώ ίδιος θα ξανάρθουμε σε αυτή την Επιτροπή για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Περιμένω πραγματικά με ανυπομονησία έναν επικοδομητικό διάλογο για την απαλλαγή που αφορά το δημοσιονομικό έτος 2010. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βεβαιώ ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου προσβλέπει στις μαζί σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προτείνω τώρα τα μέλη της Επιτροπής να συζητήσουν αυτά που έλεγχαν. Διαδραστικό, παρακαλώ. Μάλιστα, Πρόεδρε. Μια που οι περισσότερες από τις διδασκαλίες γίνονται ευθύνη των κρατών μελών, δεν θα ήταν καλό να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να κάνει τα πρώτα του σχόλια. Looks a logical uh, request. Λογικό φαίνεται το έτοιμά Εγώ δεν διαφωνώ, αλλά είναι κανένα πάνω από το Συμβούλιο. Θα με εξέπλητε. I do not see anybody. Δεν βλέπω κανένα. Οπότε δεν μπορώ να ακολουθήσω το έτοιμά σα. Θα το έχουμε κατά νου. Η κυρία Γιάννη Σέντα, διαδικαστικό επίση. Ναι. μπορούμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να είναι παρόν τουλάχιστον στην παρουσία στην Ολομέλεια. Ναι, πολύ καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα. Θα ζητήσουμε από το Συμβούλιο να είναι παρόν στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ για την πρόταση αυτή. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Τορμασία. Τώρα θα πρότεινα να δώσουμε το λόγο. Πρώτα, στον εισηγητή για την απαλλαγή του προπολισμού 2010 και μετά που θα ακούσουμε αυτά τα σχόλια και τις ενδεχόμενες ερωτήσεις μπορεί να απαντήσει η Επιτροπή και το Συνέδριο για στο τις ερωτήσεις αυτής του εισηγητή και μετά πολιτικές ομάδες και όποιος θέλει να υποβάλει ερωτήσεις. Αν συμφωνείτε θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Φιέλμαν. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Καλτέρα και τον κύριο Σεμέτα και τις παρεμβάσεις τους. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε στη σωστή προοπτική να απαλλαγή αυτού του έτους, γιατί υπάρχουν πολλές πολιτικές διαφορές. Γιατί τι γίνεται παραδείγματος σε άλλους τομείς, πολίτες, ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι παράλληλο με αυτό που κάνουμε εδώ. Ο το πιστοτικός ε, κανονισμός και είναι ετήσια περίοδος και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να συμβάλλει σε αυτές τις άλλες διαδικασίες. Πιο σημαντικό επίσης είναι να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίση εμπιστοσύνης για τον προπολογισμό και την δημοσιονομική διαχείριση των ε, πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να ξαναδημιουργήσουμε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνη που υπήρχε. Θα πρέπει να βασιστούμε σε καλή συνεργασία με την Επιτροπή και πιο σημαντικό ακόμα, μια που η κρίση αυτή εξοπιστίας βρίσκεται στα κράτη-μέλη, εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε και είναι σωματικά τα σχόλια που έκανε ο κύριος Φαγκάνη και η κυρία Αιάλα Σέντερ. Θα πρέπει να έχουμε συνεργασία των κρατών μελών. Και καταδεμεσμένη ευθύνη δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευθύνη στο ένα μέρος των αντίον. Εγώ θα ήθελα να δημιουργήσουμε διπλή ευθύνη. Και ένα άλλο σημαντικό ε, παράγοντας είναι βέβαια το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και θα ήθελα να το συγχαρώ για μια ετήσια έκθεση που πιστεύω ότι βελτιώθηκε. Βελτιώθηκε σε διαφάνεια και δίνει τώρα πιο σημαντικές και λεπτομερείς ε, και διαφανείς ε, πληροφορίες. Εκ πρώτης όψης, γιατί δεν μπορούσα να τη μελετήσω εις βάθος, η εργασία πάνω στην έκθεση αιτησίων δραστηριοτήτων είναι νομίζω ενδυναμωμένη και θα ήθελα επίση να χαιρετήσω το νέο κεφάλαιο 8 στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Καλτέρα. Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό. Δεν αποκλείεται να έχουμε καινούριε ιδέες στο μέλλον όσον αφορά τη μεθοδολογία και την παρουσίαση που θα είναι χρήσιμα στοιχεία για μας στη μελλοντική μας εργασία. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τι συμπληρωματικές αυτέ πληροφορίε και νομίζω ότι μιλάω εξ ονόματο όλων όταν λέω ότι προσβλέπουμε στην δυνατότητα ενδελεχού μελέτη. Διαβάζοντα τι διάφορε πληροφορίε και να σα κύριε Καλτέρα, περνάει το μήνυμα πολύ ξεκάθαρα. Υπάρχει σταθερότητα, δεν υπάρχουν δραματικέ αλλαγέ. Αν υπήρχαν δραματικέ αλλαγέ, ίσω θα υπήρχε λόγο ανησυχία. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι η σταθερότητα είναι καλή, η σταθεροποίηση είναι καλή. Γιατί θυμάστε, με ορισμένα στοιχεία πέρσι δεν ήμασταν ευτυχεί. Και στα σημεία που δεν ήμασταν ευτυχεί, η στασιμότητα δεν είναι καλή. Και αν κοιτάξω τι βλέπουμε να μας ε, εντυπωσιάζει, είναι η συνοχή. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλό να μην υπάρχει πρόοδος εκεί. Τούτου λεχθέντος είμαι ικανοποιημένος με την συνεχή επιτυχία σε πολλούς τομείς. Τη δυνατότητα δηλαδή της Κομισιόν να κρατήσει παραδείγματο χάρη το ποσοστό στο 2% περίπου στην Γεωργία. Είναι σημαντικό αυτό. Και εκπλήττομαι ότι το ποσοστό για τις εξωτερικές πολιτικές έχει πέσει κάτω από το 2% από την πρώτη φορά. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι προσωρινές και τελικές πληρωμές θα πρέπει να γίνονται σε υψηλότερα ποσοστά. Και αυτές είναι νομίζω, κατά τη γνώμη μου, οι πληρωμές που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τομέας της συνοχής είναι εκείνος που θα πρέπει να εξεταστεί φέτος, για να μην πω φέτος ξανά. Όταν εξέτασα το κείμενο, ε, εξέτασα καταρχήν τα χρώματα. Δεν βρήκα ακόμα τίποτα έγχρωμο. Και πήρα τα δικά μου τα χρωματιστά μου και ζωγράφισα, αν θέλετε, το κείμενο. Για να δω τι θα γινόταν αν είχατε χρησιμοποιήσει ε, χρησιμοποιήσει χρώματα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος βέβαια που έχουμε ακριβή στοιχεία τώρα και όχι χρώματα. Ε, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν ε, έχετε πια στη σημεία έγχρωμα όπου περνάει το σύστημα πολύ πιο γρήγορα. Και κοιτάξτε πώς ήταν τώρα όταν δει κανένας σε διάφορες ομάδες πολιτικών. Η εικόνα χρώμη είναι ίδια από το παρελθόν, ίσως λίγο παραπάνω πράσινο. Αλλά είναι δύσκολο να κάνει κανένα τη σύγκριση, το καταλαβαίνω, το είπατε και εσείς στην ομιλία σας, είναι δύσκολο να κάνει κανένα τη σύγκριση από έτος σε έτος. Αλλά αν δούμε τις συνολικές πληρωμές και δούμε πόσα είναι κίτρινα, πόσα κόκκινα, πόσα πράσινα. Και βλέπουμε ότι έχουμε Περισσότερο ε, πράσινα. Από 8% στο 20% περάσαμε. Πολύ καλό νέο. Αλλά έχουμε και πιο πολλά κόκκινα. Από 30% στα 33%. Και νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε αυτές τις εικόνες έτσι. Αλλά θα ήθελα να, να ακούσω γιατί δεν χρησιμοποιείται πια αυτά τα χρώματα που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε και τα ψάχνουμε τώρα. Αλλά αφήνοντα τα γενικά σχόλια κατά μέρο, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία που έτυχαν τι άμεσες προσοχή μου. Το πρώτο, η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εποπτείας. Το συνέδριο δίνει μια ανη, ε, ανητική, ε, θέση σε αυτό. Γιατί τα συστήματα ελέγχου εποπτείας δεν άπτονται παρά μόνο μερικά. Και αυτό γιατί το ποσοστό ε, σφάλματος ξεπερνάει το κατόφλι ορίμασης. Για την πολιτική συνοχή έχουμε 7,7% και τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν τα συστήματα ελέγχου εποπτείας και διαχείρισης για να είμαι σίγουρη ότι τα συστήματα λειτουργούν όπως πρέπει. Αναρωτιέμαι λοιπόν, κάνουν τα κρατημέρια αυτό που πρέπει να κάνουν. Και εκεί επανερχόμαστε πάλι στο ερώτημα που έθεσαν αρχικά οι συνάδελφοι. Εγώ θα έλεγα όχι. Στην παράγραφο 425 το λέει ξεκάθαρα το συνέδριο. Λέει εκφράζει την άποψη ότι υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες για τις αρχές των κρατών μελών για να μπορέσουν να έχουν ανοιχνεύσει και διορθώσεις τουλάχιστον κάποια από τα σφάλματα πριν προ... προωθήσουν τα στοιχεία αυτά στην Κομισιόν για 58% των συναλλαγών που έχουν επίτευξη στα σφάλματα. Είναι σημαντικό αυτό και δεν είναι καινούριο, δεν είναι επαναστατικό, αλλά παρόλα αυτά δυσάρεστο. Και το γεγονός ότι είναι, δεν είναι νέο, αλλά εξακολουθεί να είναι μέσα στο κείμενο, είναι απαράδεκτο. Κάποια κράτη-μέλη δεν μπορέσαν να διαχειριστούν τα κονδύλια ή τα σχέδια. Γιατί, γιατί ήταν πολύ πολύ πολύπλοκο, έτσι ακούμε πολλές φορές. Ή γιατί ορισμένα κράτη-μέλη δεν καταβάλουν επαρκείς προσπάθειες ή γιατί η Κομισιόν δεν έχει τα σωστά μέσα στα χέρια της για να διορθώσει. Γιατί όλες οι αλλαγές αυτές σπανίως οδηγούν σε πραγματικές απώλειες. Και αυτό είναι κάτι που αναφέρεται στην έκθεση. Ότι σπάνια, σπανιότατα οδηγούν αυτά σε πραγματικές απώλειες. Πρόκειται για μια αντίδραση του Συμβουλίου όταν υιοθετήθηκε η οδηγία. Τώρα όμως που συζητάμε για νέα οδηγία θα πρέπει νομίζω να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ερωτήματα. Πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες, καταβάλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να διορθώσουν ή θα πρέπει να είμαστε εμείς πολύ ε, αποφασιστικοί, να σταματήσουμε κάποια προγράμματα σε κάποια κράτη-μέρη στα οποία τα συστήματα ελέγχου της εποπτείας δεν είναι επαρκή. Ε, πολλά από αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να βρεθούν στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας απελαχής. Θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε τη βοήθεια που χρειαζόμαστε και τις απαντήσεις από την Κομισιόν αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και απαντήσεις από τα κράτη-μέλη, όπω είπαν και οι συνάδελφοι. Ποια είναι τα συστήματά του, τι έχουν κατά νου, πώς πιστεύουν ότι θα πρέπει να βοηθήσει η Κομισιόν, ποια θα είναι η δική του ευθύνη. Και γι' αυτό ζήτησα από τους συντονιστές να καλέσουν κράτη-μέλη σε αυτή την Επιτροπή και είδα διαβάζοντας ότι τρεις χώρες ξεχωρίζουν και θα έπρεπε να μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματά μας. Έχουν συμφέρον νομίζω να το κάνουν. Έχουν συμφέρον να επανέλθει η εμπιστοσύνη στις δημόσιες δαπάνες. Ταυτόχρονα θα θέλω Τίσιο την Κομισιόν, γιατί διαβάνονται στην έκθεση και την απάντηση της ε, Κομισιόν για 4,24, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Τρία κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τα περισσότερα σφάλματα. Ποια κράτη-μέλη μπορεί να μας το πει αυτό η Κομισιόν. Για να έχουμε καλό διάλογο μέσα στα πλαίσια της απαλλαγής με τα κράτη-μέλη που έχουν προφανώς προβλήματα στην αντιμετώπιση των ποσοστών σφάλματος τους. Εκτιμώ τις καλές ιδέες της Κομισιόν για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η διαχείριση των κρατών μελών. Αλλά θα πρέπει νομίζω να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας και στα κράτη-μέρη αυτά. Εγώ έκανα μία ανάλυση του κινδύνου και είδα ότι ο πολιτικός κίνδυνος δεν είναι αυτός που φανταζόμαστε. Γιατί εγώ δεν θέλω να ξεκινήσουμε άσκημα τη νέα περίοδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σεμέτα για αυτό που μας είπε, αλλά θα πρέπει νομίζω να συνεχίσουμε. Δεύτερη παρατήρηση. Τα μέσα ε, δημοσιονομικής μηχανικής. Αυτά αναφέρονται καταρχήν όσον αφορά τη νέα διατύπωση του δημοσιονομικού κανονισμού και δεύτερον στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2013 όπως λέγεται να, να αυξηθεί η επίπτωση του κοινοτικού ε, προϋπολογισμού είναι σαν αρχημία αυτό πώς θα βρει κανένας χρυσάφι από το μολύβι Η δική μου προκαταρκτική ανάλυση είναι η εξή. Καταρχήν υπήρχε ένα πρόβλημα λογιστικής όσον αφορά αυτό το μηχανισμό. Θα πρέπει να, συγχαρεί να συγχαρούμε την Κομισιόν που βρήκε τη λύση για το θέμα αυτό της ε, λογιστικής. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι η πραγματικότητα που κρύβεται κάτω από αυτά. Στο κεφάλαιο 4. Αυτά που διαβάζω με ανησυχούν, με φοβίζουν. Καταρχήν, τα μέσα για την περίοδο 2007-2013 αξιολογούνται στα 8,1 δις ευρώ. Σημαντικότατο ποσό. Ταυτόχρονα η παρουσία των στοιχείων από τα κράτη-μέλη προ την Κομισιόν είναι, για να μην πούμε τίποτα άλλο, ανεπαρκή. Το λέει αυτό η Κομισιόν στο σημείο 31 και 32. Αναγκάζεται η Κομισιόν να στείλει εκατοντάδε επιστολών στι διάφορε υπηρεσίε των κρατών μελών, ούτω ώστε να δώσουν τι πληροφορίε που χρειάζεται για να προετοιμάσει στους, ε, Δεν ξέρω κατά πόσον η Κομισιόν προτίθεται να προετοιμάσει την έκθεση για την απόδοση αυτών των στοιχείων. Γιατί οι κανόνες και η νομική βάση, κατά τη γνώμη μου, είναι υπερβολικά ευέλικτοι. Και δεν πιστεύω ότι έχουν δοθεί τα σωστά κίνητρα για να έχουμε τα απαραίτητα ωφέλη από τα μέσα αυτά δημοσιονομικές ε, μηχανικές να χρησιμοποιούν τα χρήματα δηλαδή πλιστάκες. Και στο 4-4 δίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα η Κομισιόν. Το προσωρινό μου συμπέρασμα θα ήταν λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντικό πρόβλημα απόδεστος στοιχείων στον τομέα και το συνέδριο λέει ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για την αγροτική ανάπτυξη όπως αναφέρεται στο 1.31 και σε άλλους τομείς πολιτικής όπως αναφέρεται στο σημείο 1.33. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα έτσι η Κομισιόν και πώς μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο σημείο. Επίσης, αναρωτιέμαι γιατί η Κομισιόν πιστεύει ότι εδώ θα βρεθεί η λύση για την πολιετή για το πολιετή προγραμματισμό, ενώ κάπου αλλού αναφέρει ότι αυτά τα μέσα μηχανικής ε, είναι επικίνδυνα. Δεν έχουμε νομίζω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα και θα πρέπει να το κάνουμε. Και το τρίτο και τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι ο κοινωνικό προπολογισμό και η δημοσιονομική κρίση. Συμφωνώ με τον κύριο Καλτέρα ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στα κράτη-μέλη αφορά και τον προπολογισμό της Ένωσης. Και συμφωνώ μαζί σας κύριε Καλτέρα ότι υπάρχει ε, κίνδυνος κενών η, η λόγω της ε, ε, ανάγκης υποστήριξης κάποιων κρατών μελών. Υπάρχουν όμως κενά και στην κοινοβουλευτική εποπτεία. Και ομολογώ ότι υποστηρίζω έντονα το αίτημα του συνεδρίου να αυξηθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Γιατί οι κίνδυνοι που υπάρχουν είναι ανοιχτοί. Κράτη-μέλη που έχουν δυσκολίες, λέγεται, έλαβαν εγγυήσεις δανείων της τάξης των 30 δις ευρώ. Τα δύο νέα μέσα για τον ε, για, τον δημοσιονομικό, για τη δημοσιονομική υποστήριξη και για την σταθερότητα έχουν όρια 50 και 60 δις. Στον ε, προπολογισμό του 2010 είχαμε μία ε, έκθεση στον ε, χρηματοπιστωτικό κίνδυνο της τάξης των 122 δις. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα εκραγεί κάποια στιγμή, αλλά δείχνει πόσο εκτεθειμένο είναι ο προπολογισμό της Ένωσης. Και αυτό χωρίς σωστούς, ε, σωστή δημόσια υποπτία και κοινοβουλευτική υποπτία και απαλληλογήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη. Αυτά είναι τα τρία πρώτα συμπεράσματα και σκέψεις που είχα όταν διάβαζα την έκθεση. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα έχουν πολύ περισσότερα να προσθέσουν σε αυτό το τομέα. Και θα κάνουμε κάτι το πολύ ενδιαφέρον φέτος νομίζω. Μια ενδιαφέρουσα άσκηση εδώ. Και προσδοκώ να υπάρχει συνεργασία όχι μόνο όπως πάντα με το ηλεκτρικό συνέδριο και την Κομισιόν και τους συναδέλφους, αλλά φέτος και από τα κράτη-μέλη. Γιατί οι καιροί απαιτούν ευθύνη όλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. ago... Πριν λίγο καιρό υπέραψα κάποιες επιστολές και καλούσα τους υπουργούς οικονομικών των τριών κρατών μελών που αναφέρονται περισσότερο ε, και είναι περισσότερο για λάθη να έρθουν στην Επιτροπή μας. Τους έχω καλέσει λοιπόν, δεν μου έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής. Εγώ θα τους καλέσω λέει, θα τους τηλεφωνήσω λέει ο μιλητής, ο εισηγητής. Κύριε Καλδέιρα, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους και σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων που δουλεύουν στο ελεγκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ για την εμφάνιση σας. Κάθε μέρα προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα για να φέρετε εις πέρας τις ευθύνες σας ε, για την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Είπαμε που η έκθεσή μας δεν είναι τόσο έγχρωμη, τόσο χρωματιστή όσο θα θέλατε, αλλά οι πληροφορίες που σας δίνουμε φέτος, ελπίζω, ότι σας επιτρέπουν να σκίσετε τα καθήκοντά σας, να κάνετε τις δικές σας αξιολογήσεις και μια τέτοια συνεργασία πάντα την εκτιμούμε. Υπάρχει ένα ουσιαστικό λόγο, ένα ουσιαστικό θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Οι συγκρίσει με έγχρωμα γραφήματα φέτο δεν θα είχε νόημα. Γιατί οι τομείς πολιτικής που, όπου εστιάζουμε φέτος είναι διαφορετικοί από αυτούς στους οποίους εστιάζαμε πέρυσι. Ε, αφερπίν, η συνοχή. Η συνοχή παλιά δεν ήταν μαζί με την ενέργεια και τις μεταφορές. Η έρευνα δεν ήταν με τις άλλες εσωτερικές πολιτικές. Θέλουμε να συγκρίνουμε συγκρίσιμα πράγματα, λοιπόν. Υπάρχει και ένας δεύτερος ουσιαστικός λόγος που δεν έχουμε χρωμαγραφήματα. γραφήματα. Φέτος, εφαρμόσαμε την ίδια μεθοδολογία, ακόμα μια χρονιά, εφαρμόσαμε την ίδια μεθοδολογία για έκτη συναπτή χρονιά. Σας δώσαμε πολλά ποσοτικά πληροφοριακά στοιχεία και κατά 95% τα στοιχεία που σας δίνουμε είναι ακριβή. Προσπαθούμε να δίνουμε πραγματικές πληροφορίες. Αυτό προτιμούμε. Γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιες πληροφορίες θα βοηθήσουν εσάς και τα κράτη-μέλη να καταλάβουν καλύτερα την εξέλιξη των πραγμάτων. Κοιτάξτε, πρέπει να, έχετε τα, να βάλετε τα πράγματα και σε ένα σωστό πλαίσιο. Να τα δείτε με τη σωστή προοπτική τους. Γιατί η σταθερότητα, λέτε, δεν είναι καλή. Είναι καλή, δεν είναι καλή, εξαρτάται από το σημείο θετηρία και το που θέλουμε να καταλήξουμε. Το γεγονό ότι δεν δώσαμε έγχρωμα γραφήματα. Το κάναμε επίτηδε. Σα δώσαμε νούμερα ούτω ώστε να αξιολογήσετε και να μετρήσετε. Από σήμερα τις εξελίξεις και να ξέρετε πώς αλλάζουν τα πράγματα σύν το χρόνο. Τα πράγματα είναι σταθερά γιατί δημιουργούμε κάποια συστήματα για κάποια χρονική περίοδο. Τα δημιουργούμε για 7 χρόνια. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η σταθερότητα. Και αυτά τα συστήματα είναι υπεύθυνα για το πώς εφαρμόζονται όλα αυτά στα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη κάνουν αυτό που δεσμεύονται να κάνουν. Σας είπα ότι για τη συνοχή, για το 58% των περιπτώσεων που υπήρχε λάθος, τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει να υποβληθεί αίτηση αποζημίωσης, επιστροφής. Πρέπει όλοι οι υπεύθυνοι σε όλα τα επίπεδα, κυρίω τα κράτη-μέλη, πούμε στον τομέα τη πολιτική συνοχή, μέχρι να λειτουργήσουν σωστά, θα υπάρχει στασιμότητα ή σταθερότητα. Παρ' όλα αυτά, στην, ε, συνοχή, στην πολιτική συνοχή δεν υπάρχει σταθερότητα. Έχουμε μια μικρή αύξηση του ποσοστού σφάλματος. Χωρίς να αλλάζουμε ριζοσπαστικά το σύστημα, ε, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αλλά πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες. Μπορείτε να πείτε, να μου διτάξετε ότι οι κανόνες είναι περίπλοκοι, θα μπορούσαμε να είναι πιο απλοί, θα μπορούσαμε να είχαμε σχεδιάσει καλύτερα τα συστήματα. Ε, αυτό ζητούμε να γίνει στη νέα περίοδο προγραμματισμού. Και με βάση τις ε, προτάσεις της Κομισιόν θα γίνει κάτι τέτοιο. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα τώρα, αλλά μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα στο μέλλον. Φυσικά, όταν αλλάζουμε τα συστήματα, τα αποτελέσματα, ε, δεν είναι τα ίδια τα επόμενα χρόνια. Και πρέπει τις αλλαγές θα τις δούμε μετά από χρόνια. Τώρα, ας πούμε, κοιτάμε ε, το οικονομικό έτος αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλος ο κύκλος είναι 2010-2013. Δεν έχουμε ακόμα ε, δει όλα τα ωφέλη που υποτίθεται ότι θα προκύψουν από τα νέα συστήματα που υιοθετήθηκαν για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Και η Επιτροπή σας έδωσε ένα παράδειγμα. Ε, ούτως ή άλλως ε, το 2010 είχαμε την πρώτη ετήσια έκθεση για τα μέσα δημοσιονομικής, δημοσιο, ε, οικονομικής, τεχνικής. Πρέπει να τονίσουμε την απάντηση που έδωσε η Κομισιόν στη δική μας σύσταση. Με βάση την ατζέντα σας σήμερα, εξετάζεται την ε, πρόταση τροποποίησης του κανονισμού που προβλέπει ότι τα προβλήματα τα οποία είναι υπέτεια για τις καταστάσεις που ανέφερα, θα αντιμετωπιστούν. Χαίρομαι λοιπόν που προτείνονται λύσεις για προβλήματα που έχουμε εντοπίσει. Και ακριβώς γι' αυτό, σε αυτόν τον τομέα, θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αντιδρά τόσο γρήγορα. Φυσικά αυτή τη στιγμή σιωθετηθούν όλα αυτά, θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν. αν εφαρμοστούν σωστά, θα επιληθεί το πρόβλημα. Αυτό ισχύει και σε σχέση με αυτά που είπα προηγουμένως για τα συστήματα ελέγχου. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Επίσης, για την ε, άποψη που εκφράσατε για την επίπτωση της κρίσης στους λογαριασμούς μας. Έχουμε αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό δημοσιονομικής ε, σταθερότητας. Θα πρέπει αυτός ο μηχανισμός να λειτουργεί σωστά με βάση σωστό έλεγχο, δημόσιο έλεγχο και θα πρέπει επίσης μια ασφαλιστική δίκλα επιπλέον να είναι και η κοινοβουλευτική εποπτεία. Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους. αυτών των μέσων α, κινδύνους για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση αποτυπώνεται η έκθεσή του στον κίνδυνο, αποτυπώνεται στου ετήσιους λογαριασμού. Και το, το συνέδριο έλεξε τους ετήσιου λογαριασμού, Ε, σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για το Ταμείο Εγγύσεων, σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για το σύστημα ε, τρεχουσών πληρωμών ε, της Ευρωζώνης και εκτός της Ευρωζώνης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχουμε εγγύησεις από τον προϋπολογισμό. Σήμερα αυτό ο μηχανισμός της δημοσιονομικής σταθερότητας επίσης εξετάζεται ε, λόγω της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπου δεν υπάρχουν εγγύησεις από τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό, ε, εστιάζουμε εκεί. Ευχαριστώ, Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Φέλνερ για τις παρατηρήσεις του, για ο κύριο Σεμέτας. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του ότι στον τομέα της πολιτικής συνοχής το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι σαφές είπε ο ίδιος ότι το 58% των σφαλμάτων εντοπίζονται στο πρώτο επίπεδο ελέγχου, στα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το πρώτο επίπεδο ελέγχου δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Και φυσικά η Επιτροπή καταβάλει κάθε προσπάθεια σε επίπεδο κατάρτισης, ούτως ώστε αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους ελέγχους να τους ασκούν αποτελεσματικά. Υπάρχουν και ανθρώπινα προβλήματα. Οι άνθρωποι αλλάζουν, έρχονται, παρέρχονται. Υπάρχει σημαντικό πηγενέλα στο προσωπικό των κρατών μελών. Και όταν έρχονται οι καινούργοι θα πρέπει να τους ε, εκπαιδεύσουμε εκ νέου, ούτω ώστε να ξέρουν ποιες είναι οι επιλέξιμες πάνες, ώστε να ξέρουν πώς θα αναξιολογούν τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες και τα σχετικά προγράμματα, κτλ. κτλ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και συμφωνώ ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες σε επίπεδο κρατών μελών. Μου ζητήσατε να κατονομάσω τρία κράτη-μέλη όπου εμφανίζονται τα περισσότερα λάθη του 2010 στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Να, το, να πω ποια είναι. Αλλά μιλήσω και σε ευρύτερο πλαίσιο. Για το 2010 Υπάρχουν σαφώ τρεις πρωτεργάτες στα σφάλματα. Ισπανία, Ιταλία και Τσεχία. Εκεί εμφανίζονται τα δύο τρίτα των λαθών που εντοπίζει το ελεκτικό συνέδριο στο τομέα της πολιτικής συνοχής. Τα δύο τρίτα λοιπόν. 16 κράτη-μέλη ελέγχθηκαν συνολικά. Και στα τρία που σας ανέφερα εμφανίζονται τα δύο τρίτα των λαθών. Και μάλιστα εμφανίζονται σε 7 προγράμματα αυτά τα δύο τρίτα των λαθών. Επικεντρώνουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να δούμε πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση. Να αναφερθώ και στην έκθεση που ετοίμασε φέτος η Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο, η οποία έχει ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2011 και λέγεται «Ανάλυση σφαλμάτων στην πολιτική συνοχής για την χρονική περίοδο 2006-2009, δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς θα προχωρήσουμε εφ' εξής. Σε αυτή την έκθεση θα βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για την κατάσταση στα κράτη-μέλη, θα δείτε κάποιες αναλύσεις και κάποιες πίνακες όπου βλέπουμε το μερίδιο του κάθε κράτους μέλους στα συνολικά σφάλματα που εντοπίζει το ελεγκτικό συνέδριο. Είπα ότι η Ισπανία, η Ιταλία έχουν τα περισσότερα λάθη για το 2010. Το ίδιο ίσχυε και για το 2006-2009. Η Ισπανία είχε το 31% των σφαλμάτων όλων των λαθών. Στην Ιταλία είχαμε το 18% όλων των σφαλμάτων που εντόπισε το ελεκτικό συνέδριο. Και, στον, και για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και το εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτή την περίπτωση το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στην τρίτη θέση χάλκινο μετάλλιο με το 10% σφαλμάτων, των συνολικών σφαλμάτων αυτή την περίοδο. Έχω, να κάνουμε τώρα κάποιες συγκρίσεις. Έχουμε την Πολωνία, που είναι μακράν ο μεγαλύτερος δικαιούχος των διαφθορτικών ταμείων. Ο αριθμός των σφαλμάτων που την αφορούν είναι μηδέν. Μηδέν λάθη για την Πολωνία. Ενώ το Βασίλειο που παίρνει πολύ πολύ λιγότερα κονδύλια από τα διευθυντικά ταμεία, είχε το 10% των συνολικών σφαλμάτων. Φυσικά υπάρχει το θέμα της Ισπανίας και της Ιταλίας. Υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα εδώ που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά και τα ίδια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανασκουμποθούν. για τη δεύτερη παρατήρησή σας. Για τα αυτά τα μέσα οικονομικής τεχνικής. Συμφωνώ ότι αυτά τα μέσα εγείρουν κάποιους κινδύνους. Ούτως, ούτως ή άλλως και το όνομα αυτό παραπέμπει αμέσως σε κινδύνους συνδέεται με κινδύνους. Σε ό,τι αφορά τη συλλογή των πληροφοριών, όπως πολύ σωστά είπατε, συλλέγουμε πληροφορίε. και το 2010 συλλέξαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια πληροφορίε και τα κράτη-μέλη ευγενώ ανταποκρίθηκαν στα αιτήματά μας. Αμέσω μετά από αυτή την προσπάθεια υποβάλαμε τροπολογίες στην νομοθεσία, ούτω ώστε να μπορούμε να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες συστηματικά. Και έτσι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που εντόπισε το ελληνικό συνέδριο. Κατά την ε, διαδικασία της απαλλαγής του τρέχοντος έτους. Εννοείται του 2010. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να συνοψίσετε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Γιατί έχουμε ένα μακρύ κατάλογο μιλητών. Για τον έλεγχο αυτών των μέσων οικονομικής τεχνικής έχουμε μία σφαιρική μεθοδολογία ελέγχων Και στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, προτείνουμε να εισαγάγουμε συστηματικά τις αναφορές, τις εκθέσεις, τη λογοδοσία δηλαδή, για αυτά τα μέσα οικονομικής τεχνικής. Για τους μηχανισμούς ε, οικονομικής σταθερότητας, όπως είπε και ο πρόεδρος Καλδέρα, οι πληροφορίε για τις δαπάνες υπάρχουν στους ετήσιους λογαριασμούς. Η δαπάνη δεν είναι από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίζεται στο δανεισμό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πρέπει να δώσει βοήθεια στα κράτη-μέλη. Και συμφωνώ ότι πρέπει να αναλύσουμε αυτόν τον τομέα. Ενδελεχώς. Το μέσο, δηλαδή χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κλπ. Και πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας εκεί. Ευχαριστώ. Τώρα τα μέλη της Επιτροπής έχουν το λόγο. Ο κύριος Καλδέιρα σε λιγότερο από μία ώρα πρέπει να φύγει για μία συνέντευξη τύπου. Προτείνω λοιπόν κάθε βουλευτής που θέλει να πάρει το λόγο να το πει. Έχω 8 άτομα, 9 άτομα στον κατάλογο μιλητών μέχρι στιγμή. Άλλο κανείς. Υπάρχουν και πάνω από 9 παρόντε τόσο ή δεν ξέρω, ίσως. Ωραία. Κλείνω τον κατάλογο. Κάθε ομιλητή έχει στη διάθεσή του 4 λεφτά. Και εν συνεχεία, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Κομισιόν θα απαντήσουν συνολικά. Καταρχάς, η κυρία Κρέσλε, για 4 λεπτά, πρώτα οι πολιτικέ ομάδε, δηλαδή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ομολογώ ότι λυπούμεθα πάρα πολύ που δεν έχουμε τη δυνατότητα συγκρισιμότητα του τρέχοντο με το περισμένο έτο. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Γιατί περιμέναμε να έχουμε συγκρίσιμους τομείς. Γιατί έτσι έχουμε την εντύπωση ακριβώς αποφεύγεται η συγκρισιμότητα. Γιατί ας πούμε συνενώστε την ενέργεια και τη συνοχή και πόσο ψηλώνει το ποσοστό σφάλματος μόνο για την συνοχή, μόνο για τις μεταφορές και ενέργεια. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα διάφορα στοιχεία. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Χρειαζόμαστε πραγματικές ε, πληροφορίες. Ίσως και λόγω της καλής συνεργασίας με την ε, Επιτροπή οδήγησε σε αυτό. Δεν είναι καλό να προσπαθούνται να καλύψετε τις ε, κακές ειδήσει, γιατί οπωσδήποτε θα εμφανιστούν. Το δεύτερο είναι τα δημοσιονομικά μέσα. Δεν αρκεί. Να μην έχει ζητήσει ήδη μια παρουσίαση από τα κράτη-μέλη η Κομισιόν στον, οργανισμό στον ε, κανονισμό του 2000. Και αυτό που είπατε για τα δημοσιονομικά μέσα δεν είναι σωστό αυτό που είπατε. Δεν υπάρχει εδώ καμία παράγραφος που να αναφέρει πώς μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα γιατί όσον αφορά την ε, δημοσιογραφική τεχνική έχουμε θέμα δημιουργικότητας. Για το Διευθυντικό Ταμείο έχουμε 137 διαφορετικά μέσα. Και σας παρακαλώ, ποιος θα ελέγχει όλα αυτά και πότε θα μπορέσει να μας δώσει ενεργικά στοιχεία το συνέδριο. Τρίτο, πρέπει να προσέχουμε γιατί το συνέδριο δεν ε, πληρεί την επιθυμία μας να κατανομάζει τα κράτη-μέλη. Δεν όλα τα κράτη-μέλη υπεύθυνα. Ε, έχουμε μεγάλα προβλήματα με λίγα κράτη-μέλη και πολλά κράτη-μέλη που δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση. Γιατί αλλιώς ε, η, η κριτική μας δεν έχει και μεγάλο αντίκτυπο, γιατί καλύπτουμε τις χώρες που φταίνε. Ρωτώ λοιπόν, πότε μπορούμε να περιμένουμε το συνέδριο να μας δίνει τα στοιχεία για τη συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Το ζητήσαμε πριστάκι σε εκθέσεις ε, απαραγής και ε, δεν το παίρνουμε ποτέ. Μετά, υπολογισμός του σφάλματος. Είναι πολύ ωραία 1,7% είναι πολύ καλό ποσοστό σφάλματος και μπορούμε να συγχαρούμε αυτούς. Νομίζω ότι εδώ συγκρίνουμε πράγματα που δεν είναι συγκρίσιμα όταν λέμε ότι κάποιες τρίτες χώρες έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Μήπως δεν μπορούμε να δούμε το σφάλμα γιατί δεν γίνεται ο σωστός έλεγχος. Μήπως αυτό είναι το πρόβλημα γιατί στη νομική βάση δεν υπάρχει κανένας όρος για τα ταμεία αυτά. Απλώς δίνουν τα χρήματα και τελειώνει. Ε, αλλιώς εσείς πώς το εξηγείτε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ αυτές τις ερωτήσεις μας. You remain completely within the four minutes. Thank you very much. No, the, I give the floor. Ευχαριστώ. Mm. Κύριος τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρουμε κύριε Πρόεδρε Καντέλα κύριε Επιτροπέ, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πολύ καλό έργο εδώ που πήραμε στα χέρια μας από το συνέδριο. Είναι μια καλή φάση με την οποία θα διασκεδάσουμε αρκετούς μήνες και θα δούμε πώς εμείς από κοινοβουλευτικής πλευρά μπορούμε να διορθώσουμε τα σφάλματα στα οποία αναφερθήκατε. Εγώ συμφωνώ με το ποσοστά κινδύνου. Ήταν καλό να τα έχουμε όλα χρώμα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο να έχουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως τα δίνουμε αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι είναι επίτευγμα που έχουμε τώρα πια ένα αριθμητικό στοιχείο για το συνολικό σφάλμα στα πλαίσια του προπολογισμού, γιατί εδώ μπορούμε να καταμετρήσουμε πραγματικά την απόδοση της Κομισιόν Παρόζο. Πρώτη φορά έχουμε κάτι τέτοιο. Γιατί τότε που είχαμε τις δικαιολογίε που λέει δεν ξέρω τι είχε γίνει, ο προκάτοχός μου, η παλιά επιτροπή ήταν υπεύθυνη, αυτά περάσαν τώρα πια. Και θα μπορέσουμε στις διάφορες ακουράσεις να αναφερθούμε σε αυτό. Έχουμε, έχω την ίδια κριτική όπως ακούστηκε ήδη για την κατανομή σε κεφάλαια. Είναι δύσκολο να συγκρίνουμε έτσι την παλαιότερη έκθεση. Αυτή εδώ το αποτέλεσμα βέβαια είναι τώρα ότι υπάρχουν περισσότεροι πράσινοι τομείς ε, κύριε Φέλναρα. αλλά θα πρέπει να δούμε τώρα γιατί δικαιολογείται αυτό. Και Χαίρομαι που υπάρχουν πολλού τομεί όπου το σφάλμα είναι τόσο μικρό, αλλά και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για την συνοχή. Ε, ε, άκουσα μια έκθεση του ε, Γενικού Διευθυντή κ. Άννα ε, στον τομέα αυτό. Ο Διευθυντικός Διευθυντής είναι από την ίδια πόλη και μάλιστα από την ίδια συνοικία όπως και εγώ και γι' αυτό του έχω πολύ εμπιστοσύνη αλλά αναφέρεται ξεκάθαρα ότι υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις. Καταλαβαίνουμε, αλλά εάν έχουμε 5% στο κάτω τμήμα της διακύμανσης και, και αυξάνεται πάνω από το 7,7% μετά, ανησυχώ. Γιατί εκεί θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν ε, να δράσει εναντί των χωρών που παράγουν τα σφάλματα και να δράσει έντονα και να υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό δείχνει πόσο ε, σημαντικές είναι οι εθνικές δηλώσεις συμμόρφωσης. Και θα πρέπει να κινηθεί εδώ η Κομισιόν να πιέσει τα κράτη-μέλη, γιατί νομίζω τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα να απομον... έχουν μάλλον συμφέρον να απομονώσουν εκείνους που σφάλουν. Και τέλος όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέσα και τις τεχνικές, το λεγόμενο engineering. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε από κοινοβουλευτικής πλευράς οι απαιτήσει που αυτή από το Κοινοβούλιο να μην ε, καταστρέψουν την συνολική εικόνα. Θα δούμε ποιες είναι οι ιδέες από την Περιφερειακή Επιτροπή ε, και πραγματικά ανησυχώ γιατί βλέπω ότι η εισηγήτρια θέλει να υπάρχει μόνο μία σελίδα ίσως αυτό να αρκεί αν δανείσει κανένας 2.000 στο, φούρνο, στο φούρναρι για να αγοράσει ένα νέο φούρνο, αλλά για πιο πολύπλοκες ε, συμβολές, δεν αρκεί. Θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας επαρκείς πληροφορίες για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και πιο πολύπλοκα θέματα. Μία σελίδα δεν αρκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Κοντέρα, τον ε, κύριο Σεμέτα και τον ε, εισηγητή κύριο Φέλνερ. Ήταν πάρα πολύ καλά τα στοιχεία για τη Γεωργία που κρατήσαμε το σωστό επίπεδο, αλλά το ανισχυρικό είναι η επιδείνωση για την συνοχή. Το είδαμε. Ξέραμε ότι το έτος 2009 ήταν ιδιαίτερα καλό, αλλά τώρα πάλι υπάρχουν ανησυχίες. Γιατί έχουμε σφάλμα στα 99%, δηλαδή τα, το ίμιση των πληρωμών ήταν αντικείμενο σφάλματος. Είναι κακό αυτό, θα πρέπει βέβαια να στραφούμε εδώ ε, στα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Επίτροπο που τόλμησε να αναφέρει τα κράτη-μέλη αυτά. Το συνέδριο δεν το έχει κάνει αυτό, αλλά χάρηκα πολύ κύριε Σεμέτα που το είπατε και υπάρχει και το έγγραφο εργασία τη Κομισιόν 2006-2009 που αναφέρει τα σφάλματα, όχι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά και τα συγκεκριμένα σφάλματα. Γιατί η Ιταλία και η Ισπανία δεν μπορούν να μάθουν από την Πολωνία μερικά πράγματα. Είναι παραδειγματική η Πολωνία. Και η πολιτική ε, εταιρική σχέσεις μεταξύ των περιφερειών είναι νομίζω καλή και θα μπορούσαμε έτσι να βοηθηθούμε για να αποφευχθούν τα σφάλματα χαίρομαι που χρησιμοποιήσατε το μέσο της διακοπής των πληρωμών, 6,2 δισεκατομμυρία είπατε, είναι ένα μέσο αυτό για να διδάξουμε πειθαρχία στα κρατημέλη και το βλέπουμε ότι ορισμένοι που αμάθαιναν στο παρελθόν δεν υπάρχουν τώρα στον κατάλογο των αμαρτωλών. Είναι πολύ καλό αυτό. Σας ευχαριστώ που υποκύψατε στην πίεση που ασκήσαμε. Μια άλλη πτυχία δική μας του Κοινοβουλίου είναι ότι οι αιτήσει ε, εκθέσεις δράσης έχουν πια λεπτομερείς ε, πληροφορίες για την ε, δημοσιονομική εποπτεία. κάνετε, κατονομάζετε και ντροπιάζετε όπως λέμε. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και για τις επιστροφές των κρατών μελών βλέπουμε ότι τα περισσότερα κράτη έχουν επιστρέψει τα χρήματα, μια χώρα δεν το έχει κάνει ακόμα, πάλι η Ισπανία. Νέα είναι η έκθεση αξιολόγησης, δηλαδή το κεφάλαιο 8 που αξιολογεί την απόδοση της Κομισιόν, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα μπορούσε να ήταν πιο αναλυτικό το κεφάλαιο αυτό, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει. Και είναι πραγματικά ανησυχητικό αυτό που λέτε, γιατί λέτε ότι υπάρχει έλλειψη προσοχής από την υποβολή αλλά και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων εξοικονομήσεις, αποτελεσματικότητα και ούτω καθεξής. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει γιατί ακριβώς σήμερα στην εποχή οικονομικής κρίσης όπου πιέζουμε τους φορολογούμενους θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική χρήση των πόρων. Θα πρέπει να υπάρχουν σταδιακοί στόχοι και θα πρέπει να βελτιωθεί εδώ η Κομισιόν και χαίρομαι που ο εισηγητής αναφέρεται ιδιαίτερα στην ε, δημοσιονομική τεχνική ή μηχανική αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό και συγχαίρω τους πάντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα το λόγο και ο κύριος Στάζ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καλντέιρα. Να ευχαριστήσω επίσης και όλους όσους ήρθαν εδώ από πλευράς του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, δούλεψαν σκληρά, ήταν ένα δύσκολο το έργο τους και νομίζω ότι ε, άλλο να έχει ένα χρονοδιάγραμμα και άλλο το να το τηρείς όπως πρέπει. Μπράβο επομένως και ε, ίσως δεν ήρθε τώρα η ώρα ακόμα να μπούμε στις λεπτομέρειες αλλά θα πρέπει απλώς να τοποθετηθούμε πολιτικά. Ακούω να αναφέρεται η έκφραση σταθερότητα. Ε, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο σταθερή η κατάσταση και η συγκυρία, ή όχι και τόσο. Γιατί σταθερή κατάσταση πάει να πει σταθερή πορεία. Αν πάμε σταθερή πορεία όμως πάει, βουλιάξε μέσα στο μέτρο κυκλώνα. Για κοιτάξτε για τα νούμερα, τι λένε υπάρχει πρόβλημα. Το 1 τρίτο όλων των συναλλαγών περιέχουν σφάλματα. Είπαμε, είχαμε πει και για πέρσι, ε, μεταφορές, συνοχή, 40,6%. 50% αλλού είχαμε πει για περιθώριο σφάλματος 50% των συναλλαγών εμφανίζουν ε, σφάλματα 7,7% περιθώριο σφάλματος Για δε τη χρήση του 2010 θέλω να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται για μια χρονιά κατά την οποία βέβαια ξεκίνησε μια θητεία, ξεκίνησατε τη δουλειά σας το Φεβρουάριο, όμως αυτό είναι ένα καμπανάκι, προειδοποίηση για τη χρήση του 11. Διότι το 11 Είναι ουσιαστικά η πρώτη χρονιά που δουλεύετε πλήρω σαν δεύτερη επιτροπή Μπαρόζο. Άρα, ρίξτε μια ματιά στα νούμερα, στα στοιχεία, αυτά που ανέφεραν οι συνάδελφοι, αυτά που είπε ο κύριο Καλτέρα. Α υποθέσουμε ότι εσεί είσαστε ένα ε, διευθυντή, ένα διαχειριστή και έπρεπε να παρουσιάσετε κάποια έκθεση για τμήματα κάποια εταιρεία. Εγώ δεν θα ήθελα στη θέση σα με τέτοια έκθεση και κυρίω, κι αν ήμουν ακόμα, δεν θα λέω ότι είναι σταθερή κατάθεση με τέτοια νούμερα. Άρα, για να κάτσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί. Όπως τα είπε ο κύριος Φιέλνερ. Τα είπε και ο κύριος Χατζημαρκάκης. Να τα συζητήσουμε. Και όταν έρθει η ώρα του απολογισμού του τι έγινε το 11, τότε να δούμε. τότε να δούμε αν η απαλλαγή θα είναι εφικτή. Επίσης, και για το Συμβούλιο είπαμε για εκείνη τη διάταξη όπου αναφέρει ότι στα πλαίσια της συνοχής και των μεταφορών έχουμε το 58% των λάθων και ο χρόνο δράση. Ε, αυτό είναι γεγονός. Η Κομισιόν τι μας λέει ότι η Τσεχία είναι υπεύθυνη για τη συντηρητική πλειοψηφία των σφαλμάτων. Να, επομένως, βασικό τμήμα της απαραίτητης μας ποιο θα είναι αυτό. Το Συμβούλιο επίσης έχει πεισματώσει. Όμως, μας το Συμβούλιο ότι δεν μπορεί στον κόσμο να λέμε τέτοια πράγματα. Εδώ μιλούμε για πάρα πολλά λεφτά. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Το Συμβούλιο, επομένω, θα πρέπει να λάβει τι ευθύνε του. Ξέρουμε τι θέλουμε, δεν χρειάζεται τώρα να μπω στι λεπτομέρειε. Αλλά, μια και πιέζει ο χρόνο, σταματώ και σα αναφέρω ότι με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω αυτά τα οποία είπε ο κύριο Φιέλνερ. Συγκεκριμένα, από την παράγραφο 34 και μετά. Διότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιου είδου παρατηρήσεις για την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου και εσύ τα είπατε κύριε Καλντέρα τα είπατε τα είπε και η Κομισιόν είπαμε για οικονομικούς ελέγχους όσον αφορά τα τεχνικά μέσα και και και πριν βάλω τελεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφο 436 είπε ότι θα διενεργήσει κάποιους οικονομικούς ελέγχους. Είναι σημαντικό να μας πείτε, Κομισιόν, πότε θα γίνουν όλα αυτά. Μην γίνει το 2015, που είπε ο κ. Καλτέρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε εμείς. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και το Ελληνικό Συνέδριο. Σας ευχαριστούμε για το λόγο. Πετέλη, ευχαριστούμε επίση και τον εισηγητή, διότι και εκείνο πάρα πολύ ξεκάθαρα τα είπε και στα συμπεράσματά του και πολλά από αυτά τα συμπεράσματα με βρίσκουν σύμφωνοι. Επίση, εγώ θα ήθελα τώρα να αναφερθώ πρώτα-πρώτα όσον αφορά το θέμα τη προχρηματοδότηση και τα σχετικά μέσα. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας τα είπε για το 2009, μας είπε τι γίνεται με αυτές τις προκαταβολές, αυτές που τώρα έχουν πάει στο ενεργητικό. Έτσι, νομίζω ότι τίθεται ένα αμφιβόλο η αξιοπιστία αυτών των λογαριασμών, διότι προδικάζουμε αυτά τα οποία διατύπωσαν οι οικονομικοί ελεγκτέ. Δεν ήταν πληρωμές, ήταν προκαταβολέ για άρα επομένω. Δεν μπορούσε τον ίδιο συνέδριο να κάτσει και να διαπιστώσει τι περιθώριο σφάλματο υπήρχε. Επομένω τώρα προβληματίζομαι, διότι εμεί είχαμε θεωρήσει ότι είναι αξιόπιστοι λογαριασμοί. Και εδώ τα έχουμε μπερδέψει. Το ηρητικό με τις ε, δαπάνες κλπ. Μιλάμε τώρα για το 50% του ενεργητικού συνολικά τέτοια ποσά, ε, άρα μιλάμε για σημαντικό ποσό και άρα σημαντικές επιπτώσεις που έχει στην αξιοπιστία. Και όπως πολλοί είπανε, φέτος το ελεγκτικό συνέδριο επέκρινε την κατάσταση σε περισσότερα από ένα σημείο μέσα στην έκθεση. Όμως δεν συμπεραίνει το συνέδριο ότι καθίστανται έτσι οι λογαριασμοί αναξιόπιστοι. Τώρα, όσον αφορά τα ταμεία Συνοχή. Το 1 του προπολογισμού είναι η συνοχή. Και εκεί έχουν 50% σφάλμα. Γιατί 50% του δείγματο είχε σφάλμα. Όμως και σε αυτή την περίπτωση δεν μας λέει το συνέδριο πού έγκυται το σφάλμα. Πόσο ουσιώδη είναι αυτά τα λάθη. γιατί θα πρέπει τότε να δούμε κατά πόσο να δώσει την περίπτωση απάντηση ή ου. Άρα θα πρέπει να μας πει ξεκάθαρα το συνέδριο τι είδου σφάλματα έχουμε για να μπορούμε και εμείς να αξιολογήσουμε την σημασία τους. Τώρα κάτι άλλο το οποίο μάθαμε από την έκθεση που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η διαφοροποίηση μεταξύ ανακτήσεων και διορθώσεων. Οι περισσότεροι μας δεν ξέρουμε ποια διαφορά υπάρχει και αυτό είναι σημαντικό. Οι ανακτήσει. είναι εκείνοι οι πόροι που παίρνονται από τους επιλέξιμους όμως οι διορθώσεις είναι χρήμα που βγαίνει από την τσέπη των φορολογουμένων άρα αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε. Δεν αναφέρονται οι διορθώσεις ούτε οι ανακτήσεις. Πόσες είναι τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν η μια ως προς την άλλη. Επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό οι διορθώσεις και ανακτήσει να αναφέρονται. Όμως είναι επίσης σημαντικό να έχουμε και προληπτική δράση, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και πότε έχουμε πρόληψη, όταν εκταμείνονται τα χρήματα για να πάνε στα κρατημέλη της Κομισιόν. Άρα, αυτό για τα κρατημέλη όμω, να μην ξεχνούμε ότι οι φορολογούμενοι στα κράτη-μέλη και όχι τα ίδια τα κράτη-μέλη τροφοδούν τον προπολογισμό και επομένω. δεν έχει σημασία, κανένας δεν νοιάζεται για ποια χώρα πρόκειται, απλώς θέλουν τα χρήματα να πιάνουν τόπο. Και κάποιος θα πρέπει να λαμβάνει την ευθύνη ότι το χρήμα πηγαίνει εκεί που πρέπει για το σωστό σκοπό. Και αν δεν υπάρχει κεντρική ευθύνη, γι' αυτό... Σας ευχαριστώ, μπορείτε να κλείσετε, λέει ο Πρόεδρος. Και κλείνω αναφέροντάς σας αυτό το οποίο ήδη αναφέρθηκε. Ακριβώς επειδή έχουμε κρίση, αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και ακριβώς λόγω της συγκυρίας κρίσης θέλω να σας πω τι έγινε με τα 60 δις που έχουν πληρωθεί ή στην Ελλάδα. στην έκθεση. Αλλά 60 δις ευρώ έχουν δοθεί στην Ελλάδα. 80 στην Ιταλία, 130 στην Ισπανία όλα αυτά δεν τα αναφέρει η έκθεση του συνεδρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ που βρισκόμαστε και θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα λεφτά πιάσαν τόπο. Ευχαριστούμε λίγο πρόεδρο. Ευχαριστούμε. Τώρα να δώσουμε το λόγο εις όσους τον έχουν ζητήσει με τη σειρά που του ζήτησαν το λόγο και πρώτη κυρία Αγιάλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα πρώτα συγχαρητήρια και ευχαριστίες ιδιαίτερες στο συνέδριο, μια που κάθε χρόνο έχουμε αυτή την έκθεση και αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε την κατάσταση των δημοσιονομικών. Να είναι επομένω πιο άρτιος ο προπολογισμό από κάθε άποψη, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεται εδώ για τις συναλλαγές και όλα αυτά να είναι διάφανα, να είναι ορατά, να τα βλέπουν οι Ευρωπαίοι. Τι είναι με τα λεφτά, πού είναι τα σφάλματα, πού είναι τα προβλήματα. Άλλο που θέλω να πω ή τον εισηγητή που τον ευχαριστώ για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Μας μίλησε για το ότι θα πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών ε, όσον αφορά την απαλλαγή, όσον αφορά την τροποποίηση του προπολογισμού, αλλά αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε επίπεδο κρατών μελών. Σε Ιρλανδία, σε Γερμανία, 55 δις εκεί, 3 δις στην Ιρλανδία. Τι γίνεται. Όλα αυτά δεν βοηθάνε στο να έχουμε εμπιστοσύνη Άρα ευτυχώ που έχουμε τώρα υπεράνω όλων το συνέδριο. Και μας λέει τι γίνεται και έτσι ξέρει ο Ευρωπαίος που πάνε τα χρήματα. Είναι σημαντικό ακριβώς μια που τώρα έχουμε δύσκολους καιρούς. Τώρα, ερώτηση προς το συνέδριο. Σε σχέση με την δεύτερη παράγραφο, συνοχή, ενέργεια, μεταφορές. Κύριε Καλτέιρο, είπατε ότι εδώ πέρα υπήρχε συγκρισιμότητα για να τα πείτε όλα αυτά. Για πέστε μας, μέσα στη συγκρισιμότητα αυτή η συνοχή εντάσσεται στην συνυπευθυνότητα ενώ ενέργεια και μεταφορές που είναι πολιτικές μας και πάρα πολύ είναι ευρωπαϊκή κυρίως αρμοδιότητα και λιγότερο κρατών μελών. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Για τη συνοχή τώρα. Που είναι μια πολιτική που μας προβληματίζει. Γιατί εδώ πέρα είπατε ότι υπάρχει αυξητική τάση για τα σφάλματα. Τι να κάνουμε για να εξηγιάνουμε τους ελέγχους της Κομισιόν. Μια από τα κράτη-μέλη πριν προβούν σε αιτήσει επιστροφών δεν κάνουν ελέγχου Τι να κάνουμε και πω θα αποφύγουμε που αυτό το πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά την πολιτική τη έρευνα που μας μιλήσατε, είπαμε ότι έχουμε περίπου το 30% συχνότητα λαθών και ε, αυτό ξεπερνάει και τη Γεωργία, βρίσκεται στη δεύτερη θέση των λαθών. Πάντω εδώ νομίζω ότι τα σφάλματα ε, είναι σχεδόν τα ίδια που ισχύουν και για τα λάθη της συνοχής. και εσείς προσφύγατε στους ανεξάρτητους οικονομικούς ελεγκτές που είναι και κάπως της μόδας. Εκεί βασιστήκατε και εμείς βασιζόμαστε για να μπορούμε να δούμε τι γίνεται από πλευράς κομισιών, από πλευράς και εδώ είχαμε 33 περιπτώσεις ε, σημαντικών λαθών, από τα οποία ήταν ακόμη πιο σημαντικά τα 14. Έρευνα και ανάπτυξη. Μιλούμε ότι από εκεί θα βρούμε τη διέξοδο για την κρίση. Άρα γι' αυτό και τα φαινόμενα των λαθών εδώ είναι σημαντικά. Ναι, ναι, πρόεδρε, θα κλείσω. Για πέστε μας τώρα τι γίνεται με τις διοικητικές δαπάνες. Πού πάει αυτό, για ποιο όργανο, για ποιο θεσμικό όργανο. Κομισιόν, για πέστε μας τώρα για την Πολωνία. Μπορείτε να κλείσετε, ο Πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι, με αυτό, με αυτό θα κλείσω, Πρόεδρε. Είναι σημαντική ερώτηση προ την Κομισιόν, γιατί μα μίλησε ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν ότι στην περίπτωση τη Πολωνία είχαμε 0% για την άξιση 9 και 10 όσον αφορά τα λάθη. Τι γίνεται με τα ποσοστά εκτέλεση για Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία συγκριτικά και πίσω για τι διοικητικέ δαπάνε, μα είπατε ότι Δεκέμβριο του 2010 φτιάξαμε την ε, εξωτερική υπηρεσία και όσον αφορά εδώ τα διοικητικά. Μπορείτε να κλείσετε, λέει ο πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι, ναι βεβαίω. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι για όλα αυτά είναι υπεύθυνη να μα απαντήσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Μακαβέη. Ευχαριστώ. Είμαι συγγήτρια για την απαλλαγή του 2010 ε, των Ευρωπαϊκών Οργανισμών. θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτά τα θέματα. Στου Ευρωπαϊκού Οργανισμού, λοιπόν. Καταρχά μα έστειλε τέτοια ετήσια έκθεση για του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι στι περισσότερε περιπτώσει, στις περισσότερε δηλαδή στους περισσότερους οργανισμούς, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από πλευρά ελεγκτικού συνεδρίου για την διαχείριση, τι προμήθειε, του ανθρώπινου πόρου, τι επιδόσει. Κανένα σχόλιο. Ουδέν. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο εμείς που είμαστε η αρχή απαλλαγής. Πώς θα λειτουργήσουμε χωρίς αυτές τις πληροφορίες. Στην περσινή έκθεση υπήρχαν τέτοια σχόλια για τις, τους οργανισμούς, για τις, τις δημόσιες προμήθειες, τα δημοσιονομικά, δημοσιονομική διαχείριση. Πέρυσι ζητήσαμε περισσότερε πληροφορίε από αυτέ που μα δώσατε και μα δίνετε λιγότερε φέτο. Σε ορισμένε περιπτώσει δεν υπάρχουν καθόλου πληροφορίε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Και ακόμα πιο σημαντικό από το γιατί είναι ότι σα ζητήσαμε να μας στείλετε αυτέ τι πληροφορίε για κάθε οργανισμό. Δεύτερο μου σχόλιο για την ειδική έκθεση για το benchmarking και την σύγκρουση συμφερόντων στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Πότε θα τα έχουμε αυτά τα στοιχεία για την έκθεση του benchmarking, ελπίζω πριν από το τέλος του 2011 και για την έκθεση που αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων πριν από το Φεβρουάριο του 2012. Αυτό ήταν ε, αυτό που είχαμε πει αρχικά. Αυτό προβλεπόταν. Θέλω να μου επιβεβαιώσετε ότι θα τηρήσετε αυτές τις προθεσμίες. Τρίτον, Χρειαζόμαστε μια ειδική έκθεση για τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότητα στις ευρωπαϊκές αυτές οι υπηρεσίες, αυτούς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ούτε καν τέσσερα λεπτά. Μπράβο. Ο επόμενος μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Καλντέιρα για την έκθεση, για την παρουσίαση. Ευχαριστώ τον Επίτροπο, τον κύριο Σεμέτας, για τις πρώτες απαντήσεις του επίσης. Τα τελευταία δύο χρόνια ζητάω, ρωτάω τον κύριο, τον κύριο Καλδέρα να δώσει σημασία και προσοχή στις επιδόσεις ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές δαπάνες. Χαίρομαι λοιπόν όπου στο κεφάλαιο 8 το συνέδριο για πρώτη φορά ε, δίνει σημασία α, στο τι πετύχαμε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, αυτό μπορεί να ξεκινήσει μια θαυμάσια παράδοση λοιπόν να έχουμε κάθε χρόνο αυτό το κεφάλαιο 8 και να το επεκτείνετε κιόλας λίγο. Εξεπλάγει από τις διαδικαστικές, τακτικές απαντήσεις της Κομισιόν στις διάφορες παραγράφους ε, του κεφαλαίου 8 για την αποτελεσματικότητα των δαπανών. Νομίζω ότι είναι πιο πολιτικό το θέμα, ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί με το, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν είναι ενδιαφέρον να μας πείτε αν η Κομισιόν δεσμεύεται από τους δημοσιονομικούς κανονισμούς ή οποιονδήποτε άλλο κανονισμό μπορείτε να φανταστείτε να εξετάσει το θέμα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Σωστό, σωστά λέει η Κομισιόν ότι μέρος του προβλήματος οφείλεται στα κράτη-μέλη που δίνουν τις πληροφορίες για το τι έχουν ε, υλοποίησει με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Φυσικά εκεί πρέπει να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις. Και τώρα πάω στο δεύτερο σχόλιο μου, Πρόεδρε, το ρόλο δηλαδή των κρατών μελών. Νομίζω ότι το λάθος που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε νέους κανόνες, νέες διαδικασίες, νέα νέα κτλ. κτλ γιατί ο ρόλος των κρατών μελών είναι άσχετος από τους κανόνες και τις διαδικασίες. Νομίζω ότι απλώς επιδεικνύουν έλλειψη πολιτικής βούλησης. Το γεγονός ότι σήμερα το Συμβούλιο απουσιάζει δείχνει ότι δεν έχουν καθόλου την πολιτική βούληση. Ας μην ε, κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από τους κανόνες αυτούς και τις διαδικασίες. Το πρόβλημα είναι σε όλα τα επίπεδα. Στα κράτη-μέλη, ε, τα εθνικά κοινοβούλια αδιαφορούν πλήρω για τον τρόπο που ξοδεύονται τα ευρωπαϊκά χρήματα. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι να έρθουν τα λεφτά στη χώρα. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια επίσης δεν έχουν τα μέσα να ασχοληθούν με τις ευρωπαϊκές δαπάνες, γιατί τα ποσά είναι σχετικά μικρά. Επομένως, σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά ε, ως βοήθεια από τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, στο Συμβούλιο δεν υπάρχει η αρχή της παρέμβασης μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή, εάν δεν μιλήσεις για τα δικά μου προβλήματα και τις δικές μου βλακίες, δεν θα μιλήσω για τα δικά σου προβλήματα και τα δικά σου ε, τις δικές σου ελλείψεις. Γι' αυτό ακριβώς σε επίπεδο Συμβουλίου δεν έχει γίνει τίποτα από τα κράτη-μέλη. Μέσα στην Ευρώπη τώρα, για μας είναι αδύνατον να μιλάμε για ευθύνη των κρατών μελών, γιατί κρύβονται πίσω από το Συμβούλιο, αν είναι παρόν, και ποτέ δεν μιλάνε για συγκεκριμένα κράτη-μέλη, δεν κατονομάζουν ποτέ χώρες. Θέλω να προτείνω, λοιπόν, να προσπαθήσουμε να καλέσουμε τους Εθνικούς Υπουργούς Οικονομικών να μας εξηγήσουν τι κάνουν με τα ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά το γεγονός ότι δεν απαντάνε σε επιστολές σας, κύριε Πρόεδρε, ε, είναι αρκετά σημαντικό και μας λέει πολλά. Μπορούμε επίση να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα διαφορετικά, να το δώσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα. Και θα ήθελα να ζητήσω τον κύριο Καλντέιρα και την Κομισιόν να μα πούν αν θέλουν να οργανώσουμε μαζί με το, να οργανώσετε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια κοινή ακρόαση όπου θα καλέσουμε διάφορου υπουργού οικονομικών και θα του ζητήσουμε δημόσια να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το κοινοτικό χρήμα, το νοσιακό χρήμα και τις δαπάνες αυτές. Μόνο με αυτή τη δημοσιοποίηση θα αντιμετωπίσουμε ε, το πρόβλημα. Ε, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη ε, για όλες τις παρατυπίες, αλλά δεν μαθαίνουμε τίποτα. Ο κύριος Ήταλα. Ευχαριστώ τον Επίτροπο, τον Πρόεδρο Καλντέιρα για την παρουσίασή του. Έχω την ίδια ανησυχία με τους συναδέλφους μου είναι η πολιτική συνοχή που με απασχολεί. Να κάνω μια απλή ερώτηση. Αυτές οι συζητήσεις τις κάνουμε εδώ και χρόνια. Όλο μιλάμε για καλύτερους κανονισμούς, καλύτερους κανόνες, καλύτερη συνεργασία, καλύτερη παρακολούθηση, αλλά τίποτα δεν αλλάζει, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Αν έπρεπε να κατονομάσετε το βασικό λόγο. Γιατί αυτό το πρόβλημα επιμένει τόσα χρόνια. Ποιος θα ήταν αυτός. Είμαστε πολύ ευγενείς. Τι πρέπει να κάνουμε κάτι την άποψή σας. Πού πρέπει να εστιάσουμε. Ευχαριστώ. Ο κ. Τσενέκη, ο τελευταίος Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Στην ίδια κατάσταση είμαστε. Κάθε χρόνο, όταν συζητάμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, πρέπει να βιαστούμε, γιατί κάθε φορά έχετε αυτή την περίφημη συνέντευξη τύπου, κύριε Πρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου, ε, εσείς πρέπει να φύγετε και εμάς μας πιέζετε και τελικά η συζήτηση περιορίζεται. Εγώ δεν συμμερίζομαι την ικανοποίηση που εκφράζει το Ελεκτικό Συνέδριο. Νομίζω ότι είναι υπερβολική αυτή η αισιοδοξία, αυτή η ικανοποίηση. Υπερβολική αυτά αρέσκεια. Νομίζω ότι μιλάμε για προβλήματα που απορρέουν από την κρίση. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι έχουν όλο και λιγότερη εμπιστοσύνη απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος των ευρωπαϊκών δαπανών. Ακριβώς και λόγω της κρίσης και λόγω όλων αυτών που προαναφέραμε. Επίσης, πρέπει να υπάρξουν μεγαλύτερες μεγαλύτερη προσπάθεια διόρθωση των, των λαθών, των σφαλμάτων. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, όπως είπε και η κυρία Ανδρέασεν, είναι σημαντικό να δούμε τι έγινε με τις ενισχύσεις που δόθηκαν ε, στην Ελλάδα. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Είναι όμως μια χώρα που είναι στην, σε πολύ ψηλή θέση, στην τέταρτη θέση παγκοσμίως, ό,τι αφορά α, για στρατιωτικές δαπάνες. Η Ελλάδα ξοδεύει το 4% του ΑΕΠ για τους εξοπλισμούς. Είναι ρεκόρ αυτό. Είπατε ότι στην Πολωνία που είναι η χώρα μου το ποσοστό των σφαλμάτων είναι 0. Ίσως αληθεύει αυτό, αλλά η αντίληψη του κόσμου στην Πολωνία είναι τελείως διαφορετική. Στην Πολωνία λέμε ότι κάνουμε συνέχεια λάθη, κυρίως σε ό,τι αφορά τα, τις δαπάνες των ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων, από τα ευρωπαϊκά ταμεία δηλαδή. Ίσως αυτή η πληροφορία του ελεγκτικού συνεδρίου ε, είναι σωστή και απλώς ε, ίσως εμείς επαναλαμβάνουμε κάποια στερεότυπα. Ή σας ξεγελάσαμε από κάποιες εκθέσεις, όπως συμβαίνει και στο παρελθόν από τις στατιστικές της Ελλάδας. Στο παρελθόν ε, λέγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ελλάδα πληρούσε όλα τα κριτήρια για να μπει στην Ευρωζώνη. Αλλά όπως ε, ανακαλύψαμε εκ των υστέρων, αυτά τα δεδομένα ήταν εσφαλμένα. Επίσης, λέτε ότι υπάρχει αλήθεια, λέμε μάλλον ότι υπάρχει η αλήθεια, η, η μισοαλήθεια, οι μισοψέματα και τα στατιστικά στοιχεία είναι το τρίτο επίπεδο. Επίσης συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλερ. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος των χρημάτων που φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πηγαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην Αφρική. Εγώ έχω πάει πολλές φορές στην Αφρική και με εκπλήσει λιγάκι το αποτέλεσμα της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου για το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου, εν συνεχεία στον επίτροπο και τέλος στον εισηγητή για να συνοψίσει. Κύριε Καλτέιρα. Ε, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων για όλες τις ερωτήσει που μου υποβάλλατε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τι δεδομένε τη χρονική πίεση. Θα προσπαθήσω όμως να το κάνω. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι το συνέδριο ελέγχει τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Πώς τα έσοδα και οι δαπάνες που χρηματοδοτεί ο προπολογισμό, πώς έχουν εφαρμοστεί, τη συγκεκριμένη οικονομική χρήση και με βάση τη συνθήκη η Κομισιόν είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο για την εκτέλεση και την απαλλαγή πάλι με βάση τη συνθήκη τη δίνεται στην Κομισιόν. Φυσικά η συνθήκη λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμόσουν τη συνθήκη. Όταν ρωτάτε το ελληνικό συνέδριο να κατανομάσει και να ντροπιάσει κράτη-μέλη, μην ξεχνάτε ότι ο έλεγχος του συνεδρίου ε, αφορά τον ενωσιακό προϋπολογισμό και δεν απευθύνεται συγκεκριμένα στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η υπεύθυνη για την εποπτεία και την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο στους τομείς κοινής διαχείρισης τα κράτη-μέλη εκτελούν και εκπληρώνουν τις ευθύνες τους για να ε, εκτελέσουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας δίνει πλήρες πληροφορίες, όχι μόνο για τις λίγες περιπτώσεις των παραδειγμάτων ή των δειγμάτων, εμείς ελέγχουμε δειγματοληπτικά τα προγράμματα στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει την ευθύνη για την εποπτεία των συστημάτων ελέγχου ελέγχει όλα τα προγράμματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Εμεί ελέγχουμε δειγματοληπτικά. Επομένως, απευθυνθείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σας δώσει όλα αυτά τα αποτελέσματα, όλε αυτές τις πληροφορίε που ζητάτε. Η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που δίδεται προς την Επιτροπή σας και προς το Κοινοβούλιο σας δίνει περισσότερες πληροφορίες για ειδικές περιπτώσεις σε εξειδικευμένα κράτη-μέλη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες εποχές που ζούμε αμφιβάλλω αν ζητήσουμε να προσλάβουμε περισσότερο προσωπικό για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα μας ε, το επιτρέψουν. Θα μας πούν όχι, αποκλείεται, δεν, ε, δεν μπορούμε να τους χρηματοδοτήσουμε. Επομένως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πιο αποτελεσματικό μπορούμε με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω περισσότερες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χρόνο με χρόνο, κύριε Γκρέσλερ. Και οι συνάδελφοί σα το είπαν, το είπα και εγώ. Έχουμε αλλάξει πολιτικέ, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσει. Δυστυχώ ότι δεν μπορώ να σα δώσω περισσότερα στοιχεία σύγκριση. Είναι αδύνατον. Μπορείτε να συγκρίνετε μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο, πενταετία α πούμε, για να δείτε συνολικά πώς εξελίχθηκε η εκτέλεση του προπολογισμού. Και στο βαθμό που υπάρχει σύγκριση, ε, σας δίνουμε παραδείγματα ε, για μια συγκεκριμένη πολιτική. Ας πούμε για την ε, συνοχή, για την γεωργία, για την έρευνα, ε, για την ενέργεια και τις μεταφορές που την βάλαμε στο ίδιο πακέτο με την πολιτική συνοχής. Αν πάτε στο σημείο 24, πάρτημα 4.1 της ετήσιας έκθεσης, μπορούμε να δούμε πόσες συναλλαγές για την ενέργεια και τις μεταφορές έχουν ελεγχθεί. Που υπάρχει συχνότητα λαθών και ποιες είναι οι επιπτώσεις στο, συνολικό ποσοστό σφαλμάτων και η σημασία. Από 8 συναλλαγές που έχουν ελεγχθεί, το 37% ήταν αλάνθαστες. Κάντε τους υπόλοιπους λογαριασμούς. Στα είχαν προβλήματα, είχαν σφάλματα. Αυτά τα λέω για να σας θέσω το πλαίσιο, να σας υπενθυμίσω ότι σας δίνουμε περισσότερες πληροφορίες, λεπτομερείς πληροφορίες που σας επιτρέπουν να κάνετε μια καλύτερη σύγκριση μέσα σε μια συγκεκριμένη όμως χρονική περίοδο. Αυτό κάνει η έκθεσή μας. Η κυρία Γκρέστερ μίλησε για τις συγκρίσεις και ότι το μαλλί το τα πάει καλύτερα από τα κράτη-μέλη. Στην εξωτερική βοήθεια, ας πούμε. Αν διαβάσατε προσεκτικά το κεφάλαιο, εγώ δεν μπορώ τώρα να μπω σε αυτό, στη δεύτερη παράγραφο του κεφαλαίου αυτού, της εξωτερικής βοήθειας, λέμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών ήταν προκαταβολές στα πλαίσια της προχρηματοδότησης. Και αν πάτε στην τελευταία παράγραφη, παράγραφο καταλήγουμε ότι οι ενδιάμεσες ε, πληρωμές και οι τελικές πληρωμές που γίνονται στο τέλος, αυτές αντιμετωπίζουν περισσότερους κινδύνους. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Του χρόνου ή στο μέλλον μπορούμε να έχουμε ε, σοβαρά προβλήματα στην εξωτερική βοήθεια και στην έρευνα και στις εσωτερικές πολιτικές. Φέτος τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι, με βάση τη γματοληψία που κάναμε και με βάση ένα σοβαρό έλεγχο, με βάση μια μεθοδολογία που εκπώνησαν κάποιοι επαγγελματίες ελεγκτές. Εκεί εντοπίσαμε λοιπόν κάποιους κινδύνους και εκεί ε, εστιάσαμε. Τώρα, λάθη. Τι λάθη έχουμε στην, ε, στην πολιτική συνοχή. Ε, δεν σέβω τους κανόνες ε, των δημοσίων προμηθειών. δεν σέβω τα, κριτήρια επιλεξιμότητας. Για να βελτιώσετε τα, τα, βασικά προβλήματα εδώ, είναι απλό. Εφαρμόστε σωστά τους νόμους των περί κρατικών προμηθειών. Δίνουμε διάφορα παραδείγματα τεχνητών διαιρέσεων των συμβάσεων, ούτω ώστε να, αποφευθούν, ή να αποφευθεί η εφαρμογή των κανόνων περί δημοσίων προμηθειών. Γίνεται αυτό στα κράτη-μέλη. Δίνουμε παραδείγματα projects, προγραμμάτων, που δεν είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση. Και παρόλα αυτά συγχρηματοδοτούνται. Τι άλλο να σας πούμε για να σε ενημερώσουμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ακόμα πιο σαφείς, να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, ούτω ώστε να εκτελέσετε κι εσείς καλύτερα τα καθήκοντά σας. Το θέμα της προχρηματοδότησης και των λογαριασμών. Εμείς θεωρούμε ότι οι λογαριασμοί παρουσιάζουν τη θέση την κατάσταση μάλλον των, ε, την οικονομική κατάσταση στο τέλος του χρόνου. Και η κάθε χρήση ε, κάνουμε τους αιτήσιους λογαριασμούς ανεξάρτητα από την προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε πολύ σημαντική, σημαντικά η προχρηματοδότηση, το αναφέρουμε και πιστεύουμε ότι με τα νέα μέσα που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αφορούν τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να εφαρμοστούν σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή αυτά τα προβλήματα για την προχρηματοδότηση θα επιληθούν. Γιατί δεν βελτιώνται τα πράγματα, ρωτάει ο κύριος Ιταλά. Το έχω απαντήσει νομίζω σε προηγούμενη ε, απάντηση που έδωσα προς τον κύριο Σίλβα. Στις σημερινές συνθήκες μπορούμε μόνο να βελτιωθούμε αν κάθε ένας από τους φορείς, κάθε δηλαδή μία από τις παραμέτρους, παίξει το ρόλο της. Ε, με βάση το σύστημα που έχουμε επιλέξει. Αλλά ε, για την επόμενη περίοδο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές. Με τον δημοσιονομικό κανονισμό θα προσπαθήσουμε και εσείς επίσης έχετε ευθύνη α, ως Επιτροπή αρμόδια που θα συζητήσει αυτόν τον κανονισμό. Ε, για να κινηθούμε προς σωστή κατεύθυνση. Να δούμε τι θα προκύψει στο τέλος των διαπραγματεύσεων. Οι νέοι κανονισμοί για τη γεωργία, για τα διαφορετικά ταμεία. Υπάρχουν. Η κυρία Γκρέσλερ μίλησε για το θέμα των μέσων ε, χρηματοοικονομικής ε, τεχνικής. Ε, ευχαριστούμε την προσοχή και προτείνουμε συγκεκριμένε λύσεις στον δημοσιονομικό κανονισμό όταν θα έχουμε το νέο ε, δημοσιονομικό κανονισμό, θα έχουμε και τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους ελεγκτές ε, να παίξουν το ρόλο του στρατιώτη, ε, ο οποίος πηγαίνει προς τον τραυματία και αγγίζει την πληγή για να δει αν όντως τραυματίστηκε. Έπειτα, μια, μια ερώτηση που έγινε για τις, τους οργανισμούς. τις agencies. Πότε λέτε θα σας δώσει α, την ε, έκθεση που σου υποσχεθήκαμε. Ε, θα τη δώσουμε εμπρόθεσμα. Η προτεραιότητα μας είναι να σας δώσουμε αυτή την έκθεση πριν τις 15 Νοεμβρίου και για τις 42-43 αυτές οι υπηρεσίες, τους 42-43 οργανισμούς. Και οι πληροφορίε που λέτε ότι λείπουν υπάρχουν σε άλλες πηγές, σε άλλες ειδικέ εκθέσεις που είναι σε αυτή τη φάση σε προετοιμασία. Αυτά τα μέσα οικονομικής τεχνικής, δημοσιονομικής τεχνικής, εξετάζονται σε διαδικασία αντιπαραβολής αυτή τη στιγμή. και εξετάζουμε και τα μέσα αυτά τέτοιες τεχνικής ε, για τα για το Ταμείο Συνοχής και τα Διαθωτικά Ταμεία. Τις ερωτήσεις που δεν μπόρεσα να απαντήσω, ε, θα μπορέσω να απαντήσω. Είμαι έτοιμος να τις απαντήσω, αν επιθυμείτε, γραπτός. Αυτά από πλευρά μου. Τώρα, λέει θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν και αν μπορείτε, κύριε Πίτροπε, να είστε σύντομος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι το γενικό επίπεδο σφάλματος είναι 3,7%. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 96% του προεπιλογισμού είναι χωρίς σφάλμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε και θεωρώ ότι οι συστήματα που εισάγονται εδώ έχουν ήδη οδηγήσει αποτελέσματα. υπάρχουν και κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία για τη συνοχή. Και θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Το επίπεδο σφάλματος στη συνοχή για το 2010 ήταν 7,7%. Αναφέρεται αυτό ρητά στην έκθεση του συνεδρίου. και τα υψηλά στοιχεία που ανέφεραν ορισμένοι οι βουλευτέ, αναφέρονται στη συχνότητα σφάλματος, όχι στο ύψο του σφάλματος. Η διαδικασία απαλλαγή ε, αυτού του έτος θα συγκεντρωθεί πολύ στην εφαρμογή των προγραμμάτων στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να προσθέσω και ο συνάδελφος Γιωάννης αν νομίζω ότι είναι έτοιμος να σας παρουσιάσει την σχετική έκθεση σε απάντηση προς τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Και τα μέλη της Επιτροπής σας μπορούν να πάρουν πάρα πολλές πληροφορίες. Και αυτό απαντάει και στην ερώτηση της κυρίας αλλά και άλλων μελών γιατί δίνονται στην έκθεση αυτή πολλές πληροφορίες. Και δίνεται επίσης μια σειρά μέτρων που εφήρμοσε η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες. Και θέλω να πω ότι οποιοδήποτε σφάλμα ε, ανείχνευσε το συνέδριο ή εμείς, παρακολουθείτε. Δεν ε, αφήνουμε δηλαδή κανένα σφάλμα χωρίς να του αποδώσουμε την κατάλληλη προσοχή. Και εξετάζουμε ποια είναι τα μέτρα για να διορθωθούν τα σφάλματα που έχει καταγράψει ο έλεγχος των δικών μας επιθεωρητών του συνεδρίου ή των ε, επιθεωρητών των κρατών μελών. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιστροφές και διορθώσεις, θα ήθελα να πιστεύω την προσοχή σας στο γεγονό ότι το σημείο 6 των ετήσιων λογαριασμών δίνει μια πλήρη εικόνα όσον αφορά τις ε, δημοσιονομικές αυτές διορθώσεις και ανακτήσεις. Ε, Πολλέ φορέ η Κομισιόν χρειάζεται συμπληρωματικέ πληροφορίε. Ε, εάν εσεί τώρα χρειαζόσαστε επίσης συμπληρωματικέ πληροφορίες, μπορούμε να σα δώσουμε όσα στοιχεία έχουμε στα χέρια μα σχετικά με τους ετησίου λογαριασμού. Κατ' γνώμη μου φέτος όμως δώσαμε τις πλήρες πληροφορίες, τουλάχιστον τις πληροφορίες που είναι σημαντικές για τη χορήγηση της απαλλαγής. Τέλος, εθίχε ένα άλλο θέμα, κατά πόσο το συνέδριο και εμείς ε, θα είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε κάποια ακρόαση. Εγώ ε, θα χαρώ να συμμετάσχω σε οποιοδήποτε ακρόαση για την οποία θα προσκληθώ. Είναι στο κάτω-κάτω και η υποχρεωσή μου να το κάνω. Εγώ προσωπικά δηλαδή θα συμμετάσχω σε όσες ακροάσεις χρειάζονται για να συζητηθούν τα προβλήματα και να οριστεί η διαδικασία της απαλλαγής. Και κάτι ακόμα όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Στάς για την θέση ε, ε, ε ανώτατου διευθυντή. Εγώ θα ήθελα να είμαι ανώτατος διευθυντής ε, στην εταιρεία αυτή, να μπορώ να ελέγχω όλες τις μονάδες. Ξέρετε όμως πάρα πολύ καλό ότι το 80% των πόρων δαπανούνται από τα κράτη-μέλη και έτσι εξαρτώμε λοιπόν από τη δική τους αποτελεσματικότητα και την δική τους αποτελεσματική χρήση των πόρων, τον δικό τους αποτελεσματικό έλεγχο. Βέβαια, η Κομισιόν καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μπορέσει να συμβολεύεται τα κράτη-μέλη για να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Άλλως, ε, επιβάλλονται κάποια μέσα για τη διακοπή των ε, πληρωμών μέσα τα οποία θα ενδυναμωθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο εφόσον ε, το Συμβούλιο και το Σώμα θα δεχθούν τις προτάσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής για να ολοκληρώσουμε και θα σας ευχαριστούσα να μιλήσετε για δύο λεπτά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Καλτέρα που επέστησε την προσοχή μας ε, στο θέμα των προκαταβολών. Πολλές υπάρχουν και δεν είναι τόσο ε, πολύ, δεν υπάρχουν τόσο πολύ στα σφάλματα όσο οι εκ των υστέρων πληρωμές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε όμως την ε, πραγματικότητα ως έχει, να μην ε, μένουμε προσκολλισμένοι σε αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου. Τα μέσα χρηματοπιστωτικής τεχνικής, μηχανικής. Εντάξει, έχουμε ασχοληθεί με το δημοσιονομικό κανονισμό επαρκώς και πολλά θα μπορέσουμε να ε, ωφεληθούμε από το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής για να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Μετά, ο κύριος Χατσιμανκάκης αναφέρθηκε στο θέμα της, ε, των διακοπών των πληρωμών. Πολύ καλό αυτό, θα συνεχίσουμε με τη δική σας συνεργασία. Καλές είναι οι διακοπές των πληρωμών, οι αναστολές. Απ' την άλλη μεριά, εάν ένα κράτος μάλλον κάνει όλο το ίδιο λάθος, δεν θα πρέπει να ξαναρχίσουν να συνεχίσουν. Καλή είναι δηλαδή η διακοπή για αναστολή. Αλλά αν δεν έχει διορθωθεί τίποτα, μην αρχίσετε να καταβάλλετε τα χρήματα. Μετά, βοήθεια. Θα πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά την αναπτυσσιακή βοήθεια. Οπωσδήποτε θα το προσθέσω στον κατάλογό μου των ειδικών ενδιαφερόντων. Χαίρομαι που έχουμε περισσότερο δεύτερο λεπτομερείς πληροφορίες. Είναι καλό αυτό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερες συγκρίσεις στο μέλλον. Αλλά, και συμφωνώ με την κυρία ε, Γκρέσλε, υπάρχει ένα πρόβλημα όταν αλλάζουν οι τομεί και τα κεφάλαια, γιατί έτσι δεν μπορούμε πολύ εύκολα να συγκρίνουμε. Καλό να έχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες, αλλά είναι πολύ πιο πολύπλοκο να συγκρίνουμε τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν σε αυτή την πρώτη ζήτη για την απαλλαγή 2010, ιδίως τον κύριο Καλτέρα και τον Επίτροπο και θα συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες έντονα. Ευχαριστώ πολύ. Διακόπτε συνεδρίαση για δύο λεπτά. Τρία λεπτά.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

Ladies and gentlemen, could you resume your... Κυρίες και κύριοι, ξανακαθίστε λέει ο Πρόεδρος. Okay, uh, I think we are now coming to point. Ωραία, και τώρα είμαστε στο το 5, το 6 και το 7 της μέσης διάταξης, λέει Πρόεδρος. Οπότε και εγώ σας προτείνω να κάνουμε τις ψηφορίες. Και μετά ό,τι μένει το συζητήσουμε. Συμφωνείτε. Εάν συμφωνείτε, τότε πάμε στο 5 της μέσης διάταξης. Έλεγχος όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση προς το Αφγανιστάν. Τροπολογία 1. Against. Υπέρ, κατά. Αποχές. Μία αποχή. Και εγκρίνεται τροπολογία 2. Ποιοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο κατά. δεν κρίνεται. Τροπολογία τρία, Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Η πλειοψηφία είναι κατά. Τέσσερα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ομόφωνα εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η πλειοψηφία είναι κατά. Το 6 είναι γλωσσικό θέμα και δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Πάμε στο 7 υπέρ Α, το 7 έχει αποσυρθεί. Πέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Πάλι είναι γλωσσικό θέμα. Ότι μου λένε, οπότε πάμε στο 9. Προφορική. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Προφορική που έχει προσθεθεί. Υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Amendment 11 is... θέμα. 12. Ποιοι είναι υπέρ. is against? is Μία εποχή. Επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Μία αποχή εγκρίνεται. 14. Γλωσσικό. 15 γλωσσικό. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία εποχή. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίθηκε ομόφωνα. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρασε. Δεν κρίνεται. κάνει. Γλωσσική, 20 γλωσσική, 21 επίσης, 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. 23, 24, 25, 26, 27 είναι γλωσσικές. 28. Πίνε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. 30, 31. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 32. Τι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33, 34, γλωσσικέ 35. Σε τρία μέρη. Πρώτο, πίνει υπέρ. Κατά. αποχέ Δύο κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ελεκτρονικό έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Ελεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 37. Προφορική απάλληψη τμήματος του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Π είναι υπέρ της τροπολογίας όπως έχει τώρα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. 38. Τρία τμήματα. Ναι, ναι, Εγώ θα ήθελα κάτι να διορθώσουμε. Γιατί συμφώνησαν ε, η εισηγήτρια κυρία Γιάρα Σέντερ αντί για την χωριστή ψηφοφορία να κάνουμε προφορική και το κείμενο να λέει σημαντικό τμήμα της ειρηνικής διαδικασίας και μέτρα για να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Άρα, πάμε τώρα στην τροποποίηση της αρχικής τροπολογίας Αγιάλα με την συγκατάθεσή της. Έτσι είναι τα πράγματα απλούστερα, δεν θα κάνουμε χωριστή ψηφορία. Άρα δεν θα κάνουμε χωριστή ψηφορία, λέει ο Πρόεδρος. Είσαστε υπέρ αυτής της τροπολογίας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Προφορική όπως τα λέει η λίστα ψηφορίας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τα 14, τι είναι υπέρ, 40 συγγνώμη, τι είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται με μία εποχή. Και τώρα, ομαδική ψηφοφορία, τροπολογίας της ΑΦΕΤ 1 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επί, τώρα ομαδική ψηφοφορία της Επιτροπής Ανάπτυξης. 1 έω 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Με ένα ψήφο κατά εγκρίνεται. Και όταν ψηφίσουμε για το σχέδιο της εκθέσεως συνολικά, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Πέρας. Σε Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα, ψήφισαν το σχέδιο της εκθέσεως όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον ε, κανονισμό του Συμβουλίου 1083 κάθετος του 2006 σε σχέση με την αρρωγή που πρέπει να ε, επιστραφεί και τα χρηματοοικονομικά μέσα. 1 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Με μία εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Αποχές. 4 Εγκρίνεται και πάμε στο 5 που είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Και μία ψήφο κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Με μία αποχή εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 17-1. Εγκρίνεται. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο σημείο αριθμών 6 της ημέρας της διάταξης θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Έρενχάουζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για την ανθρωπιστική βοήθεια. γνωρίζετε ίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι οι μεγαλύτεροι δωρητέ ανθρωπιστική βοήθειας. Το 2010 Το ποσό αυτό ήταν περίπου 36%, δηλαδή 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είχαμε μια έκθεση πρωτοβουλία που έλεγχε την αποτελεσματικότητα της ε, χρήσης της ανθρωπιστικής αυτοβοήθησης και αυτό προσπαθεί να κάνει αυτή η έκθεση. Υπήρχαν εκθέσεις της Επιτροπής ε, ΠΤΕΒΕ βέβαια, αλλά ο στόχος εκεί ήταν διαφορετικός. Υπήρχαν διάφορες ε, συναντήσεις με την Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων, με το Ελεκτρικό Συνέδριο, με την οργάνωση Voice που συνενώνει 80 μη κυβερνικές οργανώσεις, στο ΕΝΟΗΕ, με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, Ουνίτσοφ κλπ. Το πρώτο τμήμα της έκθεσης συγκεντρώνεται στον ε, έλεγχο και τους ε, μηχανισμούς εποπτείας και το δεύτερο τμήμα αφορά την εφαρμογή. Καταρχήν υπάρχουν και κεντρικά σημεία τοπικά, ιδίως η καταστροφή στο Πακιστάν και στην Αϊτή. Äh, η Γενική διαθεσιακό έχει μόνο έναν συντονιστικό ρόλο, δηλαδή η εφαρμογή επιτόπου εφαρμόζεται από τους εταίρους ΕΚΟ. η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΙΕ και άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως το Νερθρό Σταυρό. Το 39% πηγαίνει στον ΟΗΕ, το 11% στις άλλες οργανώσεις. Οι μηχανισμοί ελέγχου όσον αφορά τις κυβερνικές οργανώσεις, όσον αφορά στην ΕΚΟ και συνεργασία με τις μη κυβερνικές οργανώσεις, έχω να πω ότι υπάρχει πολύ υψηλό ποσό εργοδοσίας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια αναθεώρηση για το 2012 τη συμφωνία FPA και θα πρέπει να εξε... εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να πετύχουμε πρόοδο. Το μεγαλύτερο τμήμα του προβλήματος βρίσκεται στην ΟΗΕ που έχει την αρχή της ενιαίας, του ενιαίου λογιστικού ελέγχου. Αυτό βέβαια βοηθά να αποφευχθούν διπλές ε, επικαλύψεις και έλεγχοι αλλά από την άλλη μεριά δεν δίνονται επαρκείς πληροφορίες στους δωρητές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί και ε, ο μηχανισμός ελέγχου δεν είναι επαρκής και η πρόσβαση στα έγγραμμα δεν είναι επαρκής. Παραδείγμα χάρη η πρόσβαση στις, στα έγγραφα εσωτερικού λογιστικού ελέγχου δεν επιτρέπεται από τις περισσότερες ε, υπηρεσίες του ΟΗΕ. Υπάρχει δυνατότητα από την, το λεγόμενο Παγκόσμιο Πιστιστικό Πρόγραμμα, World Food Program, που έχει τώρα υποσχεθεί να δώσει δυνατότητα πρόσβαση στην Κομισιό στα έγγραφα αυτά. Και η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και μη γραφειοκρατικά. Δεν θα πρέπει δηλαδή ο κάθε πρόσβαση του, της Ευρωπαϊκής να πρέπει να πάει μέχρι τη Νέα Υόρκη για να δει τα έγγραφα. Θα πρέπει να μπορεί να τα πάρει και ηλεκτρονικά. Δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει στον ΕΕ για την ε, πρόσβαση στα έγγραφα είναι τα αναλυτικά έγγραφα που δεν δίνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Και επίσης η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ που ξεκίνησε το 2006 μετά το σκάνδαλο με την Βόρεια Κορέα. Και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να ασκήσουν τα κράτη-μέλη η πίεση στο ΟΗΕ για να προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση. Μετά, για την εφαρμογή. Ε, το θετικό στοιχείο είναι υπάρχουν γενικά κριτήρια. Υπάρχουν όμως και αδύναμο σημεία, δηλαδή ότι δεν ε, αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο όλα τα κράτη-μέλη της ΕΧΟ δεν έχουν τους ίδιους ελέγχους. Θα πρέπει να υπάρχει μια πιο μεγάλη ομοφωνία. Ένα τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε κατευθυντήρες τιμές όσον αφορά το κόστος ενίσχυσης, δηλαδή το χρήματα που δίνονται στους εταίρους έχω είναι άμεσα αφενός και έμεσα αφετέρου. Και το έμεσο κόστος μπορεί να φτάσει μέχρι το 7% ανάλογα την μη κυβερνητική οργάνωση. Το κόστος υποστήριξης είναι το άμεσο κόστος, εν αντιθέσει προς το γραφικό κρότος και θα πρέπει να έχουμε συγκριτικές τιμέ για τα διάφορα σχέδια για να δούμε αν υπάρχει αναλογία. Και δύο-τρία λόγια για την ΑΕΤ και το Πακιστάν. Βέβαια, μεγάλες καταστροφές είναι έκτακτες ε, υποθέσεις και θα πρέπει να ε, χρηματοδοτηθούν επαρκώς. Αλλά είδαμε για την ΑΕΤ και το Πακιστάν ότι υπήρξαν παρόμοια προβλήματα, δηλαδή ανεπαρκής ε, συντονισμός μεταξύ των ε, πρεσβειών των χωρών ε, Ανεπαρκής ανάλυση των αναγκών, η... ο... μη επαρκής όπως είπαμε συντονισμός που χρηματοδοτείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν προσπαθούμε να πετύχουμε διαφάνειες πληροφορίες, ιδίως συγκεκριμένα για το Περσιάν, θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα πρόσβαση στις εκθέσεις, εκθέσεις που δεν μας εδόθη, ούτε στις οικονομικές εκθέσεις είχαμε πρόσβαση και ε, έτσι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα συγκεκριμένο για το αποτέλεσμα. και τελικά προβλέφθηκε μια επίσκεψη αντιπροσωπεία στην ΑΕΤ και θα πρέπει να ζητήσουμε πραγματικά οικονομικέ και περιγραφικέ εκθέσει να φτάσουν στα χέρια μα πριν από την επίσκεψη αυτή για να μπορούμε να υποβάλουμε τι σωστέ ερωτήσει και να πάρουμε τι σωστέ πληροφορίε. Εν κατακλείδη, γενικά θετική είναι η αξιολόγηση. Και αν είχαμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, δεν ξέρω αν θα είχα καταλήξει το ίδιο α, συμπέρασμα. Καταρχήν όμως θετική θετικό το αποτέλεσμα, αλλά για την ανθρωπιστική βοήθεια όπως και για την βοήθεια θα πρέπει να ε, συγκεντρωθούμε περισσότερο στην προληπτική δράση, να μην αντιδρούμε πάντα, πάντα σε καταστροφές, αλλά να δούμε πόσο αηφόρες είναι οι διάφορες δράσεις που εφαρμόζουν, πόσο καλή είναι η μετάβαση από την ανθρωπιστική στην αναπτυξιακή βοήθεια και όσον αφορά τις καταστροφές, ίσως το πρέπει να τονίσουμε ένα σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση, ώστε να μπορούμε ίσω κάτι να προβλέψουμε και να μην χρειάζεται πάντα να αντιδρούμε εκ των υστέρων. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να δημιουργήσουμε μια βιομηχανία μη κυβερνητικών οργανώσεων όπου δημιουργούνται νέε εξαρτήσει. Θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιούμε τις τοπικές ικανότητε. Αυτό είναι νομίζω το πιο θετικό για το μέλλον. Αυτά, τα υπόλοιπα υπάρχουν στην έκθεση. Σα ευχαριστώ για τη συνεργασία με όλε τι πολιτικές ομάδες και ευχαριστώ και ιδιαίτερα τους βοηθούς του τους Σερνή και Ινιάν που εργάστηκαν πάρα πολύ και επίση και τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βάσα. Thank you ε, Ευχαριστώ. έχω ε, μεταξύ των, κατα... των ομιλητών τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ε, δεν αποπειρώμαι να προφέρω το όνομά του. Βίτζε, να με λέτε, είναι πολύ πιο, πιο εύκολο. Uh, Ευχαριστώ τον εισηγητή για τον πολύ επικοδομητικό τρόπο εργασίας του. Ε, συναντηθήκαμε, ήταν καλές οι συναντήσεις μας. Στην αρχή ήμασταν απρόθυμοι να ασχοληθούμε πάλι με το θέμα του ΕΚΟ. Αλλά ο τομέας είναι πολύ ασταθής, το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε είναι πολύ περίπλοκο και οι συνέπειε είναι ότι δεν είναι τα πάντα τέλεια, δεν, δεν όλα προβλέψιμα και όλα προγραμματισμένα. Η έκθεση του αναγνωρίζει, αναγνωρίζει ότι προσπαθούμε να έχουμε διαφάνεια, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες, είμαστε γρήγοροι, είμαστε ευέλικτοι και όταν οι συνθήκες επιτόπου αλλάζουν και εμείς αλλάζουμε χάρη στο δίκτυο εμπειρογνωμόνων που έχουμε επιτόπου. Και όπως είπε και ο εισηγητής, είμαστε και υπεύθυνοι και λογοδοτούμε. Γιατί θα πρέπει όχι μόνο να βοηθήσουμε όσους υποφέρουν και να μειώσουμε τα βάσανα, αλλά είμαστε και διαφανείς και λογοδοτούμε. Φυσικά υπάρχουν τομείς που μπορούμε να βελτιώσουμε. Κυρίως υπάρχει ένας τομέας, η σχέση μας με τον ΟΗΕ, που μπορούμε να, τον, να τη βελτιώσουμε. Ε, εκεί πάει το 40% της χρηματοδότησής μας και η σχέση μας είναι πολύ λεπτή και ευαίσθητη γιατί θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους. Έχουμε μια συμφωνία με τον ΟΗΕ ε, και μέσα στο αυτό πλαίσιο δουλεύουμε με μεγάλη επιμέλεια μαζί τους ούτως ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να εξετάζεται και να υλοποιεί τους στόχους της. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο ΙΕ βαθμία άλλαξε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να δίδονται και στην Κομισιόν. Με αυτόν τον τρόπο δεν κάνουμε τα ίδια πράγματα σε ό,τι αφορά την επαλήθευση. Διαιρούμε τα καθήκοντά μας. Όπως είπε ο εισηγητής, η... μίλησε για προβλήματα στο παγκόσμιο πρόβλημα διατροφής. Ο ΙΕ άλλαξε τους κανόνες για να μας βοηθήσει και η UNICEF έκανε πρόσφατα το ίδιο. Και οι άλλες υπηρεσίες λοιπόν βαθμιά ελπίζουμε θα ακολουθήσουν ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και αυτές οι εκθέσεις θα δημοσιοποιούνται ένα το χρόνο. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην πληροφορία από το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί αυτό ήταν πρόβλημα στο παρελθόν, έχει επιληθεί τώρα το συνέδριο έχει πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά και αν υπάρχει κάποια παρεξήγηση, τότε η ΕΚΟ με την ε, βοήθεια της EuroPaid επίσης βοηθάει για να ξεπεραστούν αυτές οι παρεξήγησεις δυσκολίες. Μια άλλη αδυναμία που αναφέρθηκε, η ένας βελτίωση βελτίωσης, εγώ έτσι θα το έλεγα καλύτερα, είναι ότι όλοι οι εταίροι δεν έχουν όλοι καλού εσωτερικού εταίρου. Έχουμε του μεγάλου εταίρου και του μικρού. Είναι δύο τα είδη. Οι μικροί Καλά ανάγκη δεν έχουν καλού εσωτερικού ελέγχου. Αυτό του δικού μα ελέγχου λοιπόν και στι δικέ μα αξιολογήσει κάνουμε κάποιε συστάσει προ αυτού για να βελτιώσουν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου του. Μέσω τη εταιρική σχέση μα δεν λέμε απλώ στι ΜΚΟ ότι δεν τα πήγαν καλά, αλλά του λέμε να ποιοι είναι οι τομεί οι οποίοι μπορούν να βελτιωθούν, είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο λογοδοσία, σε επίπεδο εκθέσεων, προετοιμασία εκθέσεων κτλ. Οποιοδήποτε, οποιοδήποτε το θέμα βελτιώσουμε, έχουμε μια σειρά από που ετοιμάζουμε ε, μερικές φορές ε, είναι αρκετά μακροσκελή γιατί προσπαθούν να καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα και έχουμε και ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τους εταίρους μας, τους ε, γνώμονες, τους μη τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον Ερθρό Σταυρό και τον ΟΗΕ. Υπάρχουν αυτές οι διάφορες οικογένειες. Προσπαθούμε λοιπόν να φτάσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο βελτίωσης των εσωτερικών ελέγχων. Οι έλεγχοι υπάρχουν για να υπάρχει διαφάνεια λοιπόν και για να ενισχύσουν την, ε, να υπάρχει καλύτερο consultancy για τη συγκρισιμότητα που ανέφερε εκεί ο εισηγητής. Εδώ κάνουμε σοβαρούς ελέγχους. Έχουμε το έμεσο κόστος μέχρι 7% γιατί δεν θέλουμε να μπούμε σε κάθε ανθιπολεπτομέρεια. Τα μικρά, τα τελευταία κομμάτια έχουν ελεγχθεί, αλλά το 7% αφήνουμε περιθώριο στις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ούτως ώστε να μην λογοδοτούν για κάθε απίστευτα μικρό ας πούμε έξοδο και να μην τους βαραίνουμε και υπερβολικά με γραφειοκρατικό άχθος. Ο εισηγητής είπε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη. Ο Επίτροπός μου ακριβώς αυτό κάνει. Υπάρχουν ε, πολλά έγγραφα και του Οκτωβρίου για την πρόληψη των καταστροφών και την ε, προετοιμασία μας εν καταστροφών για να είμαστε πιο ανθεκτικοί και να είναι και πιο ανθεκτικοί και εταίροι μας. Έτσι το έθεσε η Επίτροπος. Επίσης προσπαθήσαμε στις διαπραγματεύσεις για το σε δημοσιονομικό πλαίσιο να εξασφαλίσουμε ότι η μετάβαση, η σύνδεση με την αναπτυξιακή βοήθεια ε, και την βοήθεια αποκατάσταση να βρεθεί στο προσκήνιο. Εμείς κάνουμε αυτή την, ε, βάζουμε εδώ την προτεραιότητα, αλλά πρέπει να το κάνουν και οι άλλοι. Είναι θέμα εκπαίδευση, είναι θέμα του πώ ε, το βλέπουν οι άλλοι και νομίζω ότι προχωράμε προ τα εκεί. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο εισηγητής είπε ότι θα πρέπει οι τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις να αναπτύξουν το δικό τους δυναμικό. Ε, πολύ επιθυμητό αυτό πολύ και ευταίο και θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά επειδή έχουμε συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης, αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλά συστήματα ελέγχου επιτόπου, που τα διαχειριζόμαστε κεντρικά. Δεν υπάρχει κατακαιρματισμός. Ε, θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερο τους μη, κυβερνητικέ οργανώσει, τις μη οργανώσεις, αλλά θα πρέπει τα συστήματα ελέγχου να τα διαχειρίζονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μόνο. Ε, θα δούμε πώς μπορούμε να τις εμπλέξουμε απλώς στην όλη διαδικασία. Ε, ευχαριστώ την, τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεση. Ε, που με τις συστάσεις και τους προβληματισμούς ε, πραγματικά θα βοηθηθεί η ΕΚΟ και μπορεί όλα αυτά να τα δεχτεί η ΕΚΟ. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος του ελεκτικού συνεδρίου θέλει να πάρει το λόγο και να σχολιάσει. Δεν έχω σχόλια ειδικά. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα όσα είπε ο Φυσικά το θέμα είναι πολύ σημαντικό για μας, θα το ξέρετε ίσως. Σε αυτή τη φάση απλώς σημαίνω ότι οι εκθέσεις ε, της UNICEF, ε, του Παγκόσμιου Προγράμματος Επισητισμού ε, και των υπολείπων ε, agencies, των υπολείπων υπηρεσιών, οι πρώτες που ανέφερα οι δύο είναι έτοιμες και οι υπόλοιπες ακολουθήσουν. Όλα αυτά εμεί θα τα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ ε, και εμεί βεβαίω από πλευρά Ελληνικού Συνεδρίου, αλλά και φαντάζομαι και οι ευρωβουλευτέ. Ευχαριστώ. Κάποιο ευρωβουλευτή θέλει να σχολιάσει. Άρα, άρα μας πείσατε κύριε Σιγητά. Έχουμε την ημερομηνία για τις α, τροπολογίες. 15 Νοεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη. 12 η ώρα. Κλείνω και αυτό το σημείο και πάω στο τελευταίο σημείο της μέσης διάταξης. Το σημείο 9. Σας αναγκαίω λοιπόν. Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής θα γίνει τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, το απόγευμα, Τετάρτη όλη μέρα, 23 μάλλον Νοεμβρίου, όλη μέρα, και Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, πάλι όλη η μέρα συνεδρίαση. Αυτά, ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη συνεδρίαση.